collègues, nous allons reprendre... Euh, Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξαναρχίσουμε τις εργασίες της Επιτροπής μας για ένα σημαντικό θέμα που είναι η φοροδιαφυγή και οι οικονομίες των απτυσσόμενων χωρών. πρώτο μας σημείο λοιπόν για απόψε ε, είναι ε, η παρουσίαση μία, μιας μελέτης όσον αφορά της, ε, την κίνηση των φορολογικών εσόδων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι ένα θέμα επί το οποίο έχω εργαστεί όπως γνωρίζετε και που βρίσκεται στην καρδιά της αναπτυξιακής πολιτικής. Ένα αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα είναι ε, ζωτική σημασία για την ανάπτυξη, γιατί συμβάλλει στην χρηματοδότηση των δημοσίων δαπανών, αλλά και στην ενίσχυση των κρατών και της χρηστής διακυβέρνησης. Ε, σίγουρα έχουν χτυπηθεί από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, καθώς και από την πτώση των τιμών των βασικών προϊόντων. Οι αναπτυσσόμενες χώρες, λοιπόν, χρειάζονται νέου ε, νέους και ουσιαστικού πόρους χρηματοδότησης. Η κινητοποίηση, λοιπόν, των φορολογικών εσόδων είναι μεγάλο διακύ σπουδαίο διακύβευμα, ιδιαίτερα για να περιοριστεί η εξάρτηση από την εξωτερική ε, βοήθεια. Η φορολογική ανεξαρτησία των νοτίων χωρών, των χωρών του Νότου, είναι μια πολλά υποσχόμενη οδός για την ανάπτυξη των χωρών αυτών. Η αφοροδιαφυγή και η φοροαπάτη ε, καταστρέφουν τις ελπίδες ανάπτυξης των χωρών αυτών καθώς αφαιρούν ένα σημαντικό κομμάτι των εσόδων τους. Το 2009 εκτιμήθηκε πως οι αναπτυσσόμενες χώρες ετησίως έχαναν 385 δις δολάρια λόγω της φοροδιαφυγής, ε, των απατών στο διασυνοριακό εμπόριο, καθώς και λόγω των φορολογικών κινήτρων που στόχο έχουν να προσελκύσουν τα επενδυτικά κεφάλαια. Δεν ξέρω αν έχουμε νέα στοιχεία για το 2014, αλλά φοβούμαι πραγματικά πως η κατάσταση ε, δεν θα έχει πολύ βελτιωθεί. Ε, θα ήθελα να γνωρίζω και να ακούσω τους συντάκτες της έκθεσης και τους δίνω αμέσως το λόγο. Μπορείτε να δείτε μεταξύ σας, κυρία Μασκάνη και κύριε Μόρ, για να, δούμε, να δείτε ποιος θα πάρει πρώτο το λόγο. Έχετε το λόγο λοιπόν. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ που μας καλέσατε σε αυτή την συνεδρίαση. Εμείς παρουσιάζουμε την μελέτη για την κινητοποίηση των φορολογικών εσόδων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Πρόκειται για ένα άλλο ένα και πιο σημαντικό θέμα που έχει λάβει μεγάλη προσοχή πρόσφατα για τους λόγους που μόλις αναφέρατε σε σχέση με την οικοδόμηση κρατικών δομών, τη πιθανά πολιτικά ωφέλη που σχετίζονται με τον εκδημοκρατισμό και την αντιπροσωπευτικότητα καθώς και την ε, στρατηγική, τη μακροπρόθεσμη στρατηγική απεξάρτησης από την εξωτερική βοήθεια. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι σχετικά γνωστά όσον αφορά τον αναπτυξιακό διάλογο διεθνώς. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι διεθνείς φορείς ασχολούνται με αυτό το τομέα και στην έκθεση μιλήσαμε για το τι γίνεται στον τομέα αυτό. Ωστόσο, Εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες όσον αφορά τα φορολογικά έσοδα. Γιατί οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν σχετικά χαμηλές, χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές. Ένας βασικός συντελεστής είναι το ΑΕΠ που είναι χαμηλός, ε, γύρω στο 10 με 20% ε, δηλαδή, ενώ στις χώρες του ΩΣΑ είναι 30% πέρα από την χαμηλή συλλογή των φορολογικών εσόδων έχουν και χαμηλή φορολογική, ε, φορολογική ε, προσπάθεια, δηλαδή ε, και αυτό είναι το μερίδιο του τι μπορεί να συλλεχθεί από φόρους σε σχέση με το τι θα έπρεπε να συλλεχθεί. Έτσι έχουμε λοιπόν κενά, φορολογικά κενά, τα οποία αναφέρουμε και στην μελέτη μας. Το φορολογικό αυτό κενό είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτό που συλλέγουν οι κυβερνήσεις και το τι θα μπορούσαν να συλλέξουν από φορολογικά έσοδα. Δεδομένων των οικονομικών συνθήκων και της κατάστασης της εθνικής οικονομίας κάθε φορά. Η ύπαρξη ενός γενικού φορολογικού κενού ή χάσματος είναι θεσπισμένη, είναι βέβαιο ότι υπάρχει. Τώρα το πόσο μεγάλο είναι αυτό το χάσμα δεν μπορεί να το πει κανείς εύκολα γιατί υπάρχει θέμα μέτρησης που σχετίζεται με τον ορισμό του δυνητικού φορολογικού, της δυνητικής φορολογικής ε, συλλογής. Είναι πολύ δύσκολο να πει κανείς πόσα θα μπορούσε να μαζέψει μια χώρα ε, στη συγκεκριμένη οικονομική και πολιτική περίσταση της εθνικής οικονομίας, αλλά είναι επίσης δύσκολο, ακόμα και αν είχαμε μια ποσοστοποίηση αυτού του φορολογικού χάσματος, θα ήταν δύσκολο να αποδώσουμε τα μεμονωμένα φορολογικά ε, κενά σε συγκεκριμένους λόγους, σε συγκεκριμένα αίτια, όπως η φοροδιαφυγή, ας πούμε. Αντί λοιπόν να αποπειραθούμε να δώσουμε ε, ποσά, προσπαθούμε να εντοπίσουμε ποια είναι τα συστατικά των φορολογικών κενών. Εντοπίζοντας τα συστατικά μπορούμε μετά να προχωρήσουμε και να προτείνουμε δράση σε διεθνές επίπεδο ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τους συγκεκριμένους περιορισμούς. Έχουμε τρεις βασικούς ε, παράγοντες λοιπόν και σχετίζονται και οι τρεις με διεθνή θέματα. Σχετίζονται λοιπόν με τη διεθνή φοροδιαφυγή και φοροαπάτη και αυτό έχει να κάνει με πολυεθνικές εταιρείες. Το άλλο έχει να κάνει με τις ε, φοροαπαλλαγές και το τρίτο με την εξόριξη. Καταρχήν να μιλήσω για τη φοροδιαφυγή λοιπόν και να κάνω μια πρώτη παρατήρηση για, και τη φοροαποφυγή. Για, την φοροαποφυγή όταν μιλάμε έχουμε μια γενική εικόνα και εκεί συμπεριλαμβάνουμε την φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή. διαφορά είναι ότι η φοροδιαφυγή σημαίνει παράνομη δραστηριότητα, ενώ η φοροαποφυγή σημαίνει εκμετάλλευση κανόνων, νόμων προ όφελο της εταιρεία κάθε φορά, όταν μιλάμε δηλαδή για διεθνείς ε, πολυεθνικές ε, εταιρείε. Πολλές φορές υπάρχει επικάλυψη, αλλά είναι σημαντικό να έχει κάνει στο μυαλό του τη διαφορά μεταξύ των δύο. Οι διεθνείς ε, όμιλοι έχουν διάφορους τρόπους για να αποφεύγουν τη φορολόγηση. Και ένας από τους συχνότερους είναι η μεταφορά των τιμολογίων, δηλαδή μεταφέρουν τα κέρδη μεταφέρουν από δικαιοδοσίες υψηλής φορολόγησης ε, τα κέρδη τους ε, σε δικαιοδοσίες χαμηλής φορολόγησης. Κάποιες φορές αυτό, αυτού του είδους η φοροαποφυγή είναι παράνομη και κάποιες φορές όχι. Εξαρτάται από το βαθμό στον οποίο διαφέρει η πραγματική τιμή από τη συγκεκριμένη. Φυσικά υπάρχουν πολλά παραθυράκια στα διεθνή φορολογικά συστήματα. Και εμείς δίνουμε κάποια παραδείγματα στην έκθεσή μας, στη μελέτη μας, καθώς και κάποιες εκτιμήσεις για το πόσο μεγάλο και πόσο βαρύ είναι αυτό το πρόβλημα. Και η ε, Εκτιμήσεις διαφέρουν ε, σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχει μια εκτίμηση ε, από τον ΩΣΑ που λέει ότι αυτά τα θέματα φοροδιαφυγής και παράνομης μετακίνησης ποσών λέει ότι είναι τρεις φορές περισσότερη μεγαλύτερη από την αναπτυξιακή βοήθεια. Και υπάρχουν δύο βασικά συζητήματα που προκύπτουν εδώ. Καταρχήν υπάρχει σχετικά χαμηλό συντονισμό σε διεθνές επίπεδο το δεύτερο είναι ότι το σύστημα περιπλέκεται διαρκώς. Κάποιες φορές το Διεθνές Φορολογικό Σύστημα δεν έχει μπορέσει να παρακολουθήσει τους αυξανόμενα περίπλοκους τρόπους με τους οποίους οι, όμιλοι μετακινούν τα κέρδη τους και αποφεύγουν τη φορολόγηση. Και αυτό είναι πρόβλημα για τις αναπτυξιόμενες χώρες όπου οι εφορίες ε, ε, είναι περιορισμένες όσον αφορά τη διοικητική τους ικανότητα και το προσωπικό τους συνήθως οι εφοριακές αρχές στις αναπτυσσόμενες χώρες έχουν λιγότερους πόρους να αφιερώσουν για να προστατεύσουν ε, τους φορολογούμενους τους από ό,τι έχουν οι πολυεθνικές εταιρείες ώστε να σχεδιάσουν ε, επιθετικά τις φορολογικές τους υποθέσεις ώστε να αποφύγουν τη φορολόγηση. Αυτό είναι πραγματικό πρόβλημα για τις αναπτυσσόμενες χώρες φυσικά. Γίνονται ενέργειες σε διεθνές επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η διεθνής κοινότητα ανταλλάσσει ε, πληροφορίες υπάρχει ατζέντα για την διάβρωση και για την μετακίνηση κερδών. Γίνονται δράσεις λοιπόν, αλλά και πάλι η φοροδιαφυγή είναι μεγάλο πρόβλημα για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό είναι το πρώτο κενό λοιπόν. Το δεύτερο κενό, η βάση περιπτώσει συντελιστή σε ολόκληρο το φορολογικό χάσμα το οποίο αναφέρουμε σχετίζεται με τις απαλλαγές. Γι' αυτό σημαίνει τα ωφέλη όσον αφορά την φορολογική μεταχείριση των εταιριών που μπαίνουν και κάνουν επενδύσεις σε κάποια χώρα. Και υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός πολλές φορές όσον αφορά τις φοροαπαλλαγές που προσφέρονται. Είναι ιδιαίτερα εκτεταμένες στις αναπτυσσόμενες χώρες, στην Αφρική ε, και διαφέρουν μεταξύ τους. Κάποιες φορές γίνονται ad hoc διαπραγματεύσεις διαπραγματεύσει κάθε φορά σε συγκεκριμένου τομεί ή ακόμα και με συγκεκριμένε εταιρείε, που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να παρακολουθήσει κανεί ακριβώ τι συμβαίνει και να το ελέγξει. Ωστόσο αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι τα στοιχεία που έχουμε, υπάρχει και ένα, μια πρόσφατη μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας την οποία αναφέρουμε στη δική μας μελέτη, όπου αυτό που λένε είναι ότι τα φορολογικά κίνητρα δεν είναι πολύ αποτελεσματικά όσον αφορά την προσέλκυση επενδυτών. Οι επενδυτές προσελκύονται περισσότερο από πράγματα όπως ένα σταθερό πολιτικό και οικονομικό κλίμα, καλές υποδομές, διαθεσιμότητα βασικών υπηρεσιών. Περισσότερο τους προσελκύουν αυτά παρά ε, τα φορολογικά κίνητρα. Αν όντως αυτό αληθεύει, τα φορολογικά κίνητρα οι φοροαπαλλαγές αποτελούν απώλεια όσον αφορά τα έσοδα, ενώ δεν δημιουργούν πολλά έσοδα. Και πάντα μιλάω με βάση τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Τα δύο πρώτα κενά που ανέφερα λοιπόν, φοροδιαφυγή για τους ε, πολυεθνικές εταιρείες και οι φοροαπαλλαγές, αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό, σημαντική ζημία όσον αφορά το χαμένο εισόδημα, χαμένα έσοδα. Και πάλι είναι δύσκολο να μετρηθούν, αλλά είναι στο φάσμα του 20-30% του, των εσόδων κάθε φορά για τις δύο αυτές περιπτώσεις. Είναι σημαντικό πόσο πολύ μεγάλη απώλεια για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Τρίτο φορολογικό χάσμα ή κενό, το οποίο εντοπίσαμε στη μελέτη μας είναι, σχετίζεται με τις εξωτερικέ βιομηχανίες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις αναπτυσσόμενες χώρες, γιατί πολλές χώρες στην Αφρική πρόσφατα ανακάλυψαν φυσικούς πόρους πολλές ε, θα ανακαλύψουν στο μέλλον. Υπάρχει δυνητικά πολύ, πολύ, πολλά έσοδα σε αυτόν τον τομέα, αλλά πολύ συχνά τα έσοδα αυτά δεν ε, μπορούν να τα πάρουν οι ίδιες οι κυβερνήσεις. Και η αντιμετώπιση είναι αναχώρα. Υπάρχει ένα, ε, ένα μείγμα από φόρους, δικαιώματα και πολύ συχνά οι συμφωνίες αυτές είναι ad hoc. Γίνεται διαπραγμάτευση άμεσα ανάμεσα στην κάθε εταιρεία και την κυβέρνηση, πράγμα που αφήνει μεγάλο πεδίο για κακοδιαχείριση και διαφθορά. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορεί η διεθνής κοινότητα να βοηθήσει εδώ και θα μπορούσαμε αυτό να το... και το αναφέρουμε στις συστάσεις μας. Ένας από αυτούς τους τρόπους είναι να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη περιφερειακών πλαισίων για την αντιμετώπιση των εταιριών στον εξωτερικό τομέα. Ο άλλος τρόπος είναι να στηριχθούν οι εφορίες στην αντιμετώπιση αυτών των εταιριών ιδιαίτερα δηλαδή με τους επενδυτές στον εξορρυκτικό τομέα. Αυτά είναι τα τρία βασικά λοιπόν φορολογικά κενά, η φοροδιαφυγή, φοροαπαλλαγές και εξορυκτικός τομέας. Αυτά τα τρία λοιπόν, αυτοί οι τρεις συντελεστές συμβάλλουν ε, στη στα χαμηλά φορολογικά έσοδα σε αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά υπάρχουν και εσωτερικοί παράγοντες. Υπάρχουν περιορισμοί οικονομικού, πολιτικού και διοικητικού τύπου να σας αναφέρω δύο όσον αφορά τις διοικητικού τύπου περιορισμούς, που είναι το προσωπικό, η ανθρώπινοι πόροι. Πολύ συχνά είναι πολύ δύσκολο για τις εφορίες να κρατήσουν το ειδικευμένο τους προσωπικό, γιατί αυτό που μπορεί να συμβεί είναι ότι οι πιο ειδικευμένοι φεύγουν και πηγαίνουν είτε σε διεθνείς οργανισμούς, είτε σε μεγάλες λογιστικές εταιρείες και είναι πολύ δύσκολο οι εθνικές εφοριακές αρχές να κρατήσουν του ειδικού του. Επίσης, ένα άλλο παράδειγμα είναι η χρήση της ψηφιοποίησης και της ε, τεχνολογίας της πληροφορικής, όπου απαιτούνται κατάλληλα συστήματα, πράγμα το οποίο δεν υπάρχει πάντοτε, αν και έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στις αναπτυσσόμενες χώρες και στις αφρικανικές χώρες. Τώρα όσον αφορά το ρόλο της Ένωσης και τις πιθανές συστάσεις ε, για δράση. Τα καλά νέα είναι ότι γίνεται πολλή δουλειά σε αυτό το τομέα και ότι προχωρεί προς τη σωστή κατεύθυνση. Όχι μόνο από την Ένωση, αλλά από τη διεθνή κοινότητα. Υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον και αυξανόμενες δραστηριότητες από διάφορους διεθνείς φορείς. μάλλον είναι καλό αυτό, με τον μόνο κίνδυνο ότι μπορεί να υπάρχει επικάλυψη και κατακαιρματισμός των δράσεων στον τομέα αυτό, αλλά εν γέννη είναι καλό το ότι δίνεται περισσότερη προσοχή στο θέμα αυτό, κυρίως διότι το μερίδιο της αναπτυξιακής βοήθειας που αφιερώνεται στην κινητοποίηση των φορολογικών εσόδων στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι ακόμα σχετικά χαμηλό. Η χρηματοδότηση δεν είναι το μόνο ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Υπάρχει το θέμα της τεχνικής βοήθειας και άλλα. Αλλά παραμένει ένα χαμηλό ποσοστό τη γενική βοήθεια. Είναι καλό λοιπόν που γίνεται δουλειά, που γίνεται προ σωστή κατεύθυνση και στην έκθεσή μας περιλαμβάνονται διάφορα παραδείγματα δράσεων τη Ένωση αλλά και διεθνών οργανισμών στον τομέα. Τώρα, για τις δικές μας συστάσεις έχουμε δύο σύνολα συστάσεων ήταν ότι δεν θέλαμε να τις αποκαλέσουμε συστάσεις γιατί στην ουσία πρόκειται για προϋποθέσεις για αποτελεσματική δράση και το άλλο είναι συστάσεις. Όσον αφορά τις προϋποθέσεις, η πρώτη και ίσως και η πιο προφανής είναι ο συντονισμός ανάμεσα στους διάφορους ε, φορείς και όχι μόνο ο συντονισμός της Ένωσης με το τι γίνεται διεθνώς, αλλά και συντονισμός εντός ε, των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και κρατών μελών. Βεβαίως υπάρχουν αρκετοί μεγάλοι διεθνείς φορείς, ΟΣΑ, ε, το Διεθνές Μεσβατικό Ταμείο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει να παίξει ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βρει ε, ένα τομέα, τον τομέα όπου θα συνεργαστεί με τις πρωτοβουλίες που υπάρχουν ε, χωρίς να επικαλύπτεται ε, η εργασία της. Δεύτερη προϋπόθεση είναι η συμμετοχή των αναπτυσσόμενων χωρών. Σε κάποια διεθνή φόρα για τη φορολογία και ιδιαίτερα αυτά που αφορούν ανταλλαγή πληροφοριών ή μετακίνηση των κερδών, οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν να παίξουν περιθωριακά ρόλο. Αυτά τα θέματα συζητώνται πολύ ανάμεσα στις προηγμένες χώρες. Κάποιες φορές οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν συμμετέχουν επαρκώς. Υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες και εντός της Ευρώπης θα μπορούσαν να επεκταθούν και να ωφελήσουν και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Μία από αυτές είναι η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την χρηστή διακυβέρνηση των φόρων, όπου δεν περιλαμβάνονται εκπρόσωποι από τις αναπτυσσόμενες χώρες, οπότε θα μπορούσε αυτό να τους ωφελήσει θα μπορούσε να είναι μια καλή πλατφόρμα και ένα καλό μέσο για καλύτερη συμμετοχή των αναπτυσσόμενων χωρών. Είναι προϋποθέσεις αυτές για την αποτελεσματική δράση. Όσον αφορά τις τρεις συστάσεις, η μία αφορά την παγκόσμια φορολογική ατζέντα που έχει προκύψει από τις ε, συνόδους G8 και G20 και πάλι έχουμε δύο τομείς, ανταλλαγή πληροφοριών και ε, βασική διάβρωση και μετακίνηση κερδών. Αυτά θα μπορούσαν να προωθηθούν με τη συμμετοχή αναπτυσσόμενων χωρών, εξασφαλίζοντας ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες θα ωφεληθούν από αυτές τις δράσεις και από την άλλη πλευρά στις ήδη τις αναπτυσσόμενες χώρες να ενισχυθούν τα Υπουργεία οι εφορίες ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτές τις διεθνείς προκλήσεις με τη σειρά τους πιο αποτελεσματικά. Δεύτερος τομέας είναι η βοήθεια και η τεχνική αρρωγή, όπου γίνονται αρκετά, αλλά μπορούν να γίνουν και περισσότερα όσον αφορά την κινητοποίηση των φορολογικών εσόδων, όσον αφορά οικονομική βοήθεια, αλλά κυρίως τεχνική βοήθεια. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου στήριξης. Οι δύο συστάσεις, πριν να περάσω στην τελευταία, είναι σημαντικές ώστε να μπορέσουμε να οθήσουμε την παγκόσμια ατζέντα στα θέματα που σχετίζονται με τη βοήθεια και την τεχνική αρρωγή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτοί οι δύο τομεί να παίξουν ένα σημαντικό, μάλλον να δείξουν ένα σημαντικό βαθμό ευθυγράμμισης και συνοχή. Από τη μια πλευρά υπάρχει η συζήτηση περί ανάπτυξης, και είναι εκεί αποδεκτό ότι είναι σημαντική η φορολογία για τις αναπτυσσόμενες χώρες και πρέπει οι δωρητές να παίξουν το ρόλο τους ώστε οι αναπτυσσόμενες χώρες να κινητοποιήσουν περισσότερο τα έσοδά τους. Και ο πολιτικός λόγος διεθνώς επίσης ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο παραμένουν ανοιχτά θέματα όσον αφορά την εφαρμογή αυτής της ατζέντα για τα θέματα παγκόσμιας φορολογία και καθώς, κα, κατά πόσο οι αναψόμενε χώρες θα ωφεληθούν και είναι επίση πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει υψηλό βαθμό ευθυγράμμιση και συνοχή ανάμεσα στην ανάγκη αύξηση των εσόδων, πράγμα το οποίο είναι αποδεκτό, και των δράσεων σε διεθνέ επίπεδο. Τρίτη και τελευταία σύσταση που τονίζουμε στην έκθεσή μας αφορά τα περιφερειακά προγράμματα. Υπάρχουν περιφερειακοί οργανισμοί που ασχολούνται με τα φορολογικά θέματα η ΤΣΑΤ για την Νότια Αφρική, η Αφρικανική Φορολογική Διοίκηση για την Αφρική. Υπάρχει το σχετικό φόρουμ. Είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξακολουθήσει να στηρίζει αυτές τις πλατφόρμες. Όχι μόνο για την καλή δικτύωση ανάμεσα στις διοικητικές, ε, ε, μάλλον στις φορολογικές αρχές, αλλά γιατί θα μπορέσουν έτσι να αναπτυχθούν περιφερειακά προγράμματα για φορολογικά ζητήματα. Για παράδειγμα, για την ανάπτυξη κοινών αρχών που θα διέπουν τις φοροαπαλλαγές, που είναι ένα από τα φορολογικά κενά που εντοπίσαμε στην μελέτη μας. Ας πούμε να υπάρχουν οροφές, πόσες φοροαπαλλαγές και πόσο εισόδημα μπορεί κανένας να χάσει και ποιες είναι οι κατευθυντήριες γραμμές σε περιφερειακό επίπεδο. Ένας άλλος τομέας όπου θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν σχετικές συμφωνίες και προγράμματα θα ήταν στον εξωτερικό τομέα και πάλι να θεσπιστούν δηλαδή περιφερειακά πλαίσια για το πώς θα φορολογηθούν τα έσοδα από τον εξωτερικό τομέα, ώστε να μην γίνονται ad hoc συμφωνίες αναπερίπτωση ανάμεσα και στην ίδια χώρα. Αυτή είναι η τρίτη σύσταση που είχα και νομίζω ότι αυτά είχα να πω για την ώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μουρ έχει κάτι να προσθέσει. Στη συζήτηση, αν χρειαστεί, θα παρέμβω κι εγώ, λέει ο κύριος Μουρ. Πρόεδρος. Ωραία. Τότε. Οι ευρωβουλευτές. Αν έχουν ερωτήσεις για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Παρακαλώ, κύριος Βένσον. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Είναι θλιβερό να ακούει κανείς το τόσο χαμηλό ποσοστό όταν ασχολούμαστε με την αποτελεσματικότητα. Μιλάμε για 385 δισεκατομμύρια, το φαντάζεστε. Νομίζω ότι θα σας ενδιέφερε να βρίσκαμε κάποια χώρα η οποία να βρίσκεται στο σωστό δρόμο, κάποια χώρα που θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι αποτελεί το πρότυπο, το μοντέλο που να δείχνει ότι αν κανείς παρέμβει με το σωστό τρόπο τότε μπορούν τα πράγματα να γίνουν καλά, δηλαδή επέλθουν οι αλλαγές που χρειάζεται. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Εγώ τότε. Γιατί και εγώ θέλω να ξέρω κατά πόσο μπορέσατε να μελετήσετε και την μεταφορά ε, όσον αφορά τις τιμές, πόσο πολύ κοστίζουν όλα αυτά στις προσανάπτυξη χώρες και να μας δίνετε κάποιο παράδειγμα χώρας που έχει αλλάξει τις ρυθμίσεις, τους κανόνες και έχει βελτιωθεί η κατάσταση όσον αφορά την ε, φοροδιαφυγή για παράδειγμα. Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα, Καρόλα Νούνες. Παρακαλώ κύριε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που καλέσατε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σχολιάσει την μελάτη τη μελέτη αυτή. Το θέμα της φορολογίας είναι ένα θέμα το οποίο παρακολουθεί στενά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και μάλιστα χάρη σε εσά ήταν ε, εφικτό να καταλήξουμε σε μια ανακοίνωση το 2010 για τη σχέση της φορολογίας με την ανάπτυξη. Και χάρη στη δικιά σας ε, την ε, στήριξη εκπονήσαμε και κατευθυντήριες γραμμές και ξεκινήσαμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή δράσεις. Για μας δύο διαστάσεις υπάρχουν όταν μιλάμε για την φορολογία και την ανάπτυξη. Η μία διάσταση έχει να κάνει με τη διμερή μας συνεργασία. Επ' αυτού προσπαθούμε να στηρίξουμε τις δομές στις χώρες μέλη, να στηρίξουμε πολιτικές μεταρρυθμίσεις και συνεργαζόμαστε στενά και με άλλους εταίρους, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Παγκόσμια Τράπεζα, διμερείς δωρητές και για να αναφερθώ σε μία από τις συστάσεις της μελέτης, υπάρχει στενός συντονισμός μεταξύ των εταίρων. Για παράδειγμα, υπάρχει το International Tax Compact και το International Tax Dialogue. Η άλλη διάσταση είναι η διεθνής διάσταση. Και εκεί είναι που τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα. Αυτό συμβαίνει επειδή εκεί συμμετέχουν διάφοροι εταίροι και επιχειρήσεις και κυβερνήσεις και βέβαια και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή, η απάτη και η φοροαποφυγή. Δεν είναι μια εύκολη διάσταση αυτή. Συνεργαζόμαστε στενά με τον ΟΣΑ, με την Παγκόσμια Τράπεζα και όσον αφορά την ε, ε, μεταφορά των τιμών έχουμε συνεργασία και με την Παγκόσμια Τράπεζα και με τον ΟΑΣΕ και έχουμε κάποια ενδιαφέροντα επιτυχή παραδείγματα. Κολομβία, Ανδούρες, ε, Παναμάς, με τη Γερμανία και την Ελβετία που έχουν συμμετάσχει σε τέτοια συνεργασία και εκεί οι τριμερείς ε, πρωτοβουλίες έφεραν αποτελέσματα. Στηρίζουμε όμως και τις περιφερειακές πρωτοβουλίες είναι και αυτή μια σύσταση της μελέτης. Και στηρίζουμε τις ε, ε, φορολογικές αρχές στην Αφρική και την Λατινική Αμερική. Συνεπώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει ενεργά. Τη σύσταση για τον συντονισμό, ναι συμφωνούμε, πιστεύουμε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, το κάνουμε όμως, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που συμμετέχουν η συμμετοχή τώρα των υποανάπτυξη χωρών. Και αυτό είναι κάτι που προσπαθούμε να πετύχουμε, δηλαδή μια μακροχρόνια συμμετοχή των ΠΕΠΣ για παράδειγμα, κάτι το οποίο εγκρίθηκε στους G20. Γνωρίζουμε όμως ότι η πλειοψηφία των αναπτυσσόμενων χωρών λείπει από εκεί. Προσπαθούμε να στηρίξουμε τη συμμετοχή τους. Έχουμε επίσης συνεργαστεί και με τα Ηνωμένα Έθνη για να υιοθετήσουμε σχετικές κατευθυντήριες γραμμές. Όσον αφορά τώρα την σχέση της τεχνικής αρρωγής και της ανάπτυξης. Και εδώ είναι θέμα πολιτικού διαλόγου. Μετά την ανακοίνωσή μας για την φορολογία και την ανάπτυξη, υπήρξαν προτάσεις που αναφέρονταν και σε αυτά τα θέματα και που τους δίνανε μεγάλη προτεραιότητα. Έχουμε επίσης και μία γραμμή streamline στον πολιτικό μας διάλογο με τους εταίρους μας και στα κριτήρια επιλεξιμότητας για την δημοσιονομική βοήθεια. Πρόκειται για δράσεις που αναλαμβάνουμε. Τέλος, υπάρχει και μια άλλη διάσταση που αναφέρθηκε όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται στενά και συμμετέχουμε στο IDI, αλλά πάμε και πέρα από αυτό, γιατί το IDI είναι μια εθελοντική πρωτοβουλία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως το έχει πει και ξαναπεί, και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την προσέγγιση αναχώρα. Πολύ σημαντικό για την διαφάνεια στην εξορυκτική βιομηχανία. Προκειμένου λοιπόν να συνεχιστεί η καρποφόρος αυτή η δουλειά. Θα έχουμε και κάποια γραπτά σχόλια, εφόσον επιθυμείτε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευχαρίστως να σας τα δώσει. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Άλλος, παρακαλώ, θέλει το λόγο. Το προσωπικό μήπως, εφόσον κάποιος θέλει να πάρει το λόγο, ευχαρίστως γιατί ξέρω ότι κάποιοι από τους συνεργάτες μας ασχολούνται με αυτά τα θέματα και ξέρουν πολλά από αυτόν. Καλώς. Ωραία, τότε θα δώσω και πάλι το λόγο στην κυρία Μασκάνη για να απαντήσει στις ερωτήσεις που ετέθηκαν και στα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ κυρία Μασκάνη. Ευχαριστώ πολύ. Θα ζητήσω από τον κύριο Μόρ που είναι εδώ μαζί μου να απαντήσει στα σχόλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να αναφερθώ στην ερώτηση του κυρίου Σβένσον για το τι είναι θετικό εδώ πέρα. Η γενική απάντηση νομίζω είναι πως υπάρχουν πολλά θετικά. Μπορώ να αναφέρω τουλάχιστον έξι χώρες αφρικανικές όπου είχαμε σοβαρές αυξήσεις ε, της ε, συλλογής των φόρων ως ποσοστό του ΑΕΠ. Επί σειρά ετών. Η Τανζανία, Μοντζαβίκη, Γκάνα, κάποια στιγμή η Ρουάντα πήγαινε καλά, η Ουγκάντα. Το Νεπάλ επίσης προσφάτως. Υπάρχουν λοιπόν πολλές θετικές περιπτώσεις, αλλά σε γενικές γραμμές η υπόθεση αυτή είναι κάτι που γίνεται αργά και βασανιστικά. Είναι δύσκολο να διατηρηθεί κάτι τέτοιο πάνω από πέντε χρόνια. Αλλά αν δούμε συνολικά το τι γίνεται σε χώρες χαμηλού εισοδήματος, δεν είναι καταστροφή. Έχουμε την τεχνολογία, ξέρουμε πως μπορούμε να αυξήσουμε τη φορολογία και υπάρχουν πάρα πολλοί ικανοί και εκπαιδευμένοι άνθρωποι στη φορολογική διοίκηση της Αφρικής. Υπάρχει καλή βάση λοιπόν. Κύρια Πρόεδρε, για το δικό σας το ερώτημα μετά για τη μεταφορά των κερδών στο εξωτερικό το πρώτη εξέλιξη είναι πάρα πολύ θετική. Ακόμα και πριν από 2-3 χρόνια ήταν πάρα πολύ συνήθες ε, να αμφισβητεί κανείς ε, το εάν το transfer pricing είναι καν σημαντικό ζήτημα. Που έρχονταν πολυεθνικές εταιρείε και έλεγαν δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πλέον όλοι δέχονται πως συμβαίνει. Είναι μια υπόθεση που υπάρχει πίσω από όλες τις μεταρρυθμίσεις. Νούμερα δεν υπάρχουν. Τα μόνα αξιόπιστα νούμερα που ξέρω είναι κάποια του Δουνουτού που αναφέρονται σε μια χώρα και λένε πως επί τη βάση της τεχνικής τους αρρωγής σε μια μη κατονομαζόμενη χώρα χαμηλού εισοδήματος υπολογίζουν πως οι απώλειες ε, από το transfer pricing ισούνται με το 20% των φορολογικών εσόδων. Σοβαρό νούμερο υποψιάζομαι πως ε, δεν θα πάει παραπέρα το δονοτού, δεν θα μας πούν εάν είναι κάτι το χαρακτηριστικό, αλλά θεωρώ πως είναι πράγματι ε, ένα νούμερο χαρακτηριστικό για τις χώρες χαμηλού εισοδήματος. Υπάρχουν λοιπόν τεράστια πιθανά ωφέλη και μας ρωτήσατε για τυχόν επιτυχίες. Υπάρχουν επιτυχίες, ε, ιδιαίτερα η Ινδία προσφάτως έχει επιτύχει μεγαλύτερη πρόοδο στην μείωση των χειρότερων ε, περιπτώσεων από αυτές, αλλά η κατηγορία μαζί με τη Βραζιλία και την Κίνα κατ' ουσίαν έχουν επιβάλει δικούς τους κανόνες στην φορολόγηση των πολυεθνικών. Δεν σκοπεύουν να ακολουθήσουν την αρχή του ΟΣΑ και κατ' ουσίαν θεωρούν πως εάν ε, οι εταιρείες τους παρουσιάζουν λογαριασμούς που δεν στέκουν όσον αφορά το τζίρο στη χώρα τους, θα επιβάλλουν τους δικούς τους κανόνες και θα, κάτι θα πρέπει να πληρώσουν οι εταιρείες. Αυτό είναι θετικό, αλλά ε, αυτές είναι εγώμενες χώρες BRICS, δηλαδή μεγάλες, ισχυρές, με ισχυρές φορολογικές διοικήσεις. Το πρόβλημα για τις μικρές φτωχές χώρες είναι πως δεν έχουν την οργάνωση και την πολιτική και οικονομική ισχύ να κάνουν κάτι τέτοιο. Και νομίζω πως από τη σκοπιά της Κομισιόν θα έπρεπε νομίζω να είμαστε ικανοποιημένοι για το ότι ο ΣΑ κάνει κάποιες προσπάθειες. Αυτοί οι οποίοι έχουν επιβάλει αυτή τη στιγμή τις μεταρρυθμίσεις είναι οι χώρες του ΟΣΑ και η Μπρικ Και όπως είπε και η συνάδελφος, οι φτωχές χώρες είναι εκτός. Και είναι πιθανόν κάποιες από αυτές τις ε, αλλαγές να μην ωφελήσουν τις περισσότερες φτωχές χώρες για καιρό. Και υπάρχουν δύο λόγοι εδώ πέρα. Ο ένας είναι πως συχνά δεν έχουν το προσωπικό και τα συστήματα για να εκμεταλλευτούν και τα όσα έχουν για να ζητήσουν π.χ. πληροφορίες από άλλες χώρες. Και το άλλο είναι πως οι απαιτήσει για να ζητήσει κανείς απευθείας ανταλλαγή πληροφοριών είναι μεγάλες και θα περάσουν χρόνια πριν ε, είναι σε θέση να κάνουν κάτι τέτοιο οι αφρικανικές χώρες. Οπότε Υπάρχουν άλλα ζητήματα που πρέπει να δούμε εντωμεταξύ μεταξύ όπως την ε, πιθανότητα για φτωχές χώρες χαμηλού εισοδήματος εμείς, δηλαδή η διεθνής κοινότητα, να μην απαιτεί αμοιβαία αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά να επιτρέψουμε στις χώρες αυτές να ζητούν πληροφορίες, να τις λαμβάνουν κατόπιν αιτήματος, αυτομάτως, ακόμα και αν δεν μπορούν να ανταποδώσουν. Ευχαριστώ. Ε, I should like Ερώτηση έχω να σας κάνω. Μας είπατε πως ε, το Δουνουτού έχει κάνει μια μελέτη για μια χώρα την οποία δεν κατονομάζει. Εντυπωσιακό αυτό. Γιατί κρύβουν το όνομα της χώρας. Και μπορείτε να μας πείτε κάτι για τη μεθοδολογία με την οποία κατέληξαν σε αυτό τον αριθμό. Δεν μπορώ να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Εάν ήταν εδώ το Δονοτού, πιστεύω, η απάντησή του θα ήταν πως ε, λάβαμε αυτές τις πληροφορίες σε εμπιστευτική βάση στο πλαίσιο μιας αποστολής τεχνικής άρωγης, οπότε θα παραβιάζαμε την εμπιστευτικότητα αν σας εξηγούσαμε το πώς λάβαμε αυτές τις πληροφορίες ή, ή ε, το όνομα της χώρας. Ε, προσωπικά, κυρία Πρόεδρε, θεωρώ πως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κάνει ε, κάτι περισσότερο. Νομίζω πως ε, είναι ένα υπονοούμενο αυτό για το ποιο θεωρούν ότι είναι ένα μέσο νούμερο. Αλλά δεν ξέρω, ίσως εσάς να απαντούσαν, εμένα δεν μου απάντησαν πάντως. Θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ, να ακούσουμε μάλλον τον κύριο Φλόριαν Κρέγκ, ο οποίος είναι εδώ πέρα και εκπροσωπεί την ECDPM. Μπορείτε να μοιραστείτε κάποιες σκέψεις μαζί μας. Uh, thank you very much, uh, Madam Chair. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους εδώ εκ δεξιών για μια πάρα πολύ χρήσιμη μελέτη. για το τι γίνεται στις ανθρώπινες χώρες. Κοιτάξτε, φαντάζομαι δεν χρειάζεται να σας πούμε ποιοι είμαστε αλλά θεωρούμε πως είναι πάρα πολύ επικαιρή στιγμή παρουσίασης αυτής της ε, μελέτης. Τώρα, εγώ όταν διάζα την έκθεση θεώρησα πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σημειώνει μόνο μεγάλη πρόοδο στην φορολογική νομοθεσία και διαφάνεια αλλά και βεβαίως ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός ε, φορέας στον τομέα αυτόν. Οπότε ναι, πρώτον ε, σημειώθηκαν, σημειώνονται μεγάλες πρόοδοι. Μόνο την προηγούμενη εβδομάδα νομίζω είχαμε μία πρόοδο όσον αφορά την ε, ιδιοκτησία των εταιριών και όπως λέει η έκθεση η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα μοντέλο ενιαίας ε, φορολογίας, τη λεγόμενη κοινή φορολογική βάση όμως είναι σημαντικό πως ε, όταν μιλάμε για την ευθυγράμμιση με τις διεθνείς πρακτικές να μην ε, ξεχνάμε και την ισχύ του παραδείγματος. Επίση, ε, ένα αποτέλεσμα είναι πως ε, τα λόμπι τα οποία κανονικά θα έρχονταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάνε σε αφρικανικές χώρες για να επηρεάσουν τους ε, πολιτικούς. Κατ' τα στοιχεία που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια είναι πως χώρες οι οποίες είχαν κάποια πρόοδο στην πολιτική αυτή, η Γκάνα και η Κένια, υφίστανται πιέσεις για να γίνουν κέντρα offshore εξωχώριων εταιριών. Και το θέμα είναι τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μετά όπως ήδη σημειώθηκε όσα σημειώνει κάποια πρόοδο αλλά είναι πρόοδος η οποία είναι πάρα πολύ γρήγορη για να μπορέσουν να ανταποκριθούν οι αναψώμενες χώρες ειδικά στον αφορά την αυτόματη ανταλλαγή προφοριών. Χτες το βράδυ έλαβα ένα email από τον ΩΣΑ που έλεγε υπερήφανα πως πάνω από 40 χώρες έχουν συνυπογράψει την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών και ε, είναι μόνο πέντε οι αναψώμενες χώρες εκεί. Και οι λόγοι νομίζω αναφέρθηκαν από τον κύριο Μούρ. Το δεύτερο που θα έλεγα επίσης αφορά τον, την ισχύ του παραδείγματος. Θα πρέπει δηλαδή να συνεχίσετε να εργάζεστε, όπως είπαν και οι συνάδελφοι από την Κομισιόν, με περιφερειακούς οργανισμούς, αλλά πέρα από αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μοντέλο περιφερειακής ολοκλήρωσης και έχει εργαστεί στο μέτωπο αυτό επιτυχώς και αργά και βασανιστικά ορισμένε φορές με τις κοινότητες αυτές. Όταν λοιπόν φτάνει κανείς στο μια τελωνιακή ένωση, κοινή αγορά, η εναρμόνιση της φορολογικής νομοθεσίας ε, έρχεται, ακολουθεί και αυτή. Τι κάνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν ε, μιλάμε π.χ. για νικητές ή καλά παραδείγματα μπορούμε να μιλήσουμε για την κοινότητα Ανατολικής Αφρικής όπου υπάρχει μια φιλοδοξία για ένα καθεστώς κοινής φορολογίας σαν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν ε, υπόδειγμα συμφωνιών αποφυγής ε, διπλής φορολογίας και στην επόμενη προγραμματική περίοδο και Νομίζω πως είναι κάτι το οποίο μπορείτε να στηρίξετε και εσείς. Τέλος, επίσης ε, για το πλαίσιο αυτό του προπολογισμού θα ήθελα να επισημάνω πως υπάρχουν κάποιοι προβληματικοί τομείς στην αναπτυξιακή βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν αναφέρονται ακριβώς στην κινητοποίηση των πόρων αυτών, αλλά σχετίζονται στενά, αλλά δυστυχώς από φαίνεται έχουν ξεχαστεί θα αναφέρω εδώ πέρα την δέσμευση για την προστασία της κοινωνικής προστασίας και των τοπικών αρχών στις αναπτυσσόμενες χώρες, κατά το οποίο βέβαια σχετίζεται με την ανάπτυξη ενός συστήματος φορολογίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρκετά μεγάλη εμπειρία στους τομείς αυτούς, αλλά τη μοιράζεται αρκετά. Νομίζω πως ε, αυτό είναι κάτι το οποίο θα δείτε τους επόμενους μήνες. Αυτά τα σχόλιά μου και αναμένω βέβαια και τη συζήτηση, τη συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ. Κυρία Μασκάνη, θέλετε να πείτε κάποια λόγια. Ναι, σας ευχαριστώ. Νομίζω πως ε, τα σχόλια ήδη τα ανέφερε ο κύριος Μουρ και ο Φλόριαν. Οπότε θα ήθελα εγώ μόνο να επανέλθω λίγο στο ζήτημα για τις εκτιμήσεις αυτές ε, των ε, παράτυπων ροών. Να σας πω πίσω κάτι. Ε, αυτά αναφέρονται βεβαίως και στη μελέτη, αλλά ενδιαφέρουν πολύ οι εκτιμήσεις. Π.χ. Ε, από την Christian Aid 2009 μιλάνε για 165 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο για το transfer pricing. Ένα άλλο νούμερο μεταξύ 660 και 870 δισεκατομμυρίων για γενικώς ε, κάποιες ε, παράνομες ροές ε, κεφαλαίων. Γι' αυτό ακριβώς ε, εμείς δεν κάναμε κάποια προσπάθεια να καταλήξουμε σε ένα νούμερο. μεγάλο το κενό και υπάρχει εδώ πέρα ρόλος ε, που μπορεί να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω πως πέρα από τις άλλες συστάσεις που ανέφερα όπως είπατε η δύναμη του παραδείγματος είναι σημαντική. Πρωτοβουλίες εντό Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες θα βοηθήσουν όχι μόνο τις ευρωπαϊκέ χώρες, αλλά και τις αναπτυσσόμενε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρουσιάσατε την μελέτη αυτή. Σας διαβεβαιώ ότι η Επιτροπή μας θα συνεχίσει να παρακολουθεί το θέμα αυτό που είναι τόσο πολύ σημαντικό για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Τώρα συνεχίζουμε και περνάμε στο σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης. Θέσεις των χωρονακές σχετικά με τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης. Είναι ένα θέμα που έρχεται και ξανάρχεται, πολύ σημαντικό όμως, στις σχέσεις μας με τους εταίρους μας από τις χώρες ΑΚΕ. Χωρίς άλλη καθυστέρηση θα δώσω το λόγο λοιπόν στους συντάκτες της μελέτης για να μας παρουσιάσουν τα κύρια σημεία της. Είναι δύο πάλι. Είναι η κυρία Αιλίν Κουά και ο κύριος Πίτερ Λούνενμπορκ. Έχετε ένα τέταρτο στη διάθεσή σας. Μπορείτε να μοιράσετε το χρόνο μεταξύ σας, εφόσον επιθυμείτε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και την Επιτροπή σας που μας προσκαλέσατε. Η μελέτη είχε να κάνει με την θέση των ε, εταίρων στις διαπραγματεύσεις με τις χώρες ΑΚΕ που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητήσαμε την άποψη των ε, παραγόντων που κάνουν τις διαπραγματεύσεις από κυβερνήσεις, βουλευτές, κοινωνία των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα. Όλοι γνωρίζετε τις λεπτομέρειες της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης, άρα δεν χρειάζεται να σας παρουσιάσω τη συμφωνία αυτή. Πρέπει όμως να σας πω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια κατάσταση διλήμματος, στην Αφρική ιδιαίτερα ανάμεσα στο άμεσο κόστος εφόσον ε, δεν υπογραφεί τέτοια συμφωνία που σημαίνει ότι χάνεται η προτίμηση και για πολλές ε, χώρες η πρόσβαση στην αγορά, η ελεύθερη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό θέμα για αυτές. Απ' την άλλη μεριά όμως, αν υπογραφεί η συμφωνία αυτή, τότε υπάρχουν προβλήματα ενδεχομένω για την εσωτερική βιομηχανία που είναι λιγότερο ανταγωνιστική απέναντι στην ευρωπαϊκή. Υπάρχει ο φόβος για το περιφερειακό εμπόριο και το εσωτερικό εμπόριο ότι επίσης θα επηρεαστεί αρνητικά γιατί τα ευρωπαϊκά προϊόντα θα μπουν μαζικά στις αφρικανικές αγορές. Κάτι το οποίο θα έχει συνέπειες και όσον αφορά την περιφερειακή ολοκλήρωση, γιατί το βασικό στοιχείο αυτής είναι οι εμπορικές σχέσεις. Πολλές αφρικανικές εξαγωγές δεν γίνονται εκτός Αφρικανικής Υπήρου, αλλά μέσα στην Αφρικανική Ήπειρο. Υπάρχει και το θέμα της ανεργίας, εφόσον υπάρξουν αρνητικές συνέπειες. Υπάρχει και το θέμα της γεωργίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε αρνηθεί να βάλει και αυτό το θέμα στο τραπέζι και οι αφρικανικές χώρες, οι αγρότες της Αφρικής ανησυχούν γιατί λένε ότι θα είναι... Ε, θα υπάρχει κίνδυνος. Θα χαθούν έσοδα. Είπανε ότι τα έσοδα από τους δασμούς είναι κάτι το οποίο χρειάζονται οι κυβερνήσεις. Άλλου είδους φορολογία μπορεί να μην είναι τόσο αποτελεσματική. Και κυρίως υπάρχει το θέμα της πρόσβασης στην αγορά αγαθών. Προκύπτουν και νέα θέματα με το δεύτερο στάδιο της οικονομικής αυτής συμφωνίας, το θέμα του, των επενδύσεων, τον ανταγωνισμό, κανόνες για την πνευματική ιδιοκτησία κλπ. Ο συνάδελφός μου, Πίτερ, θα σας μιλήσει περισσότερο για το δίλημα αυτό και για την άποψη των ε, εταίρων. Ευχαριστώ πολύ. Αν δείτε γιατί χώρες μιλάμε, μιλάμε για την ακτή Λεφαντοστού και Γκάνα πρώτα απ' όλα. Οι άμεσες συνέπειες είναι η παρουσία του στην αγορά όσον αφορά τα προϊόντα κακάο. 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια είναι εξαγωγές τους. Πρόκειται για σπόρους, αλλά πρόκειται και για ε, κρέμα κακάο και για άλλα προϊόντα κακάο. Τα προϊόντα αυτά θα υποβάλλονται σε δασμούς και σύμφωνα με κάποιους υπολογισμούς τα προϊόντα αυτά θα καταλήξουν σε 91 εκατομμύρια δολάρια δασμούς. Το μισό των δασμών αν οι χώρες αυτές ήταν στο DSP. Συγχρόνως όμως, αν διατηρήσουν τις εξαγωγές τους στην απασχόληση, γιατί υπάρχουν σημαντικές δραστηριότητες, τότε επίσης θα υπάρχει κόστος και ένα από αυτό θα είναι απώλεια εισοδήματος είναι 600 με 700 εκατομμύρια δολάρια για την Κάνα. Και αυτό λοιπόν, όταν κοιτάμε την Δυτική Αφρική, η πρόσβαση στην αγορά εξαρτάται κατά πολύ, όπως λένε οι βουλευτές, ο ιδιωτικό τομέας και η κοινωνία των πολιτών, από την συμφωνία αυτή. Έχει υπάρξει κάποια τεχνική συμφωνία στον Ντακάρ, 75% όσον αφορά τους δασμούς, αλλά από πλευράς αξία σημαίνει ελευθέρωση πάνω από 80% των εισαγωγών από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Αφρική. Αυτός είναι ένας τομέας με ιδιαίτερο δυναμικό. Η κοινωνία των πολιτών στην Κάνα, για παράδειγμα, ζήτησε από τον πρόεδρο να μην υπογράψει, ακριβώς εξαιτίας αυτού του θέματος της πρόσβασης στην αγορά. Στη Δυτική Αφρική λοιπόν, η κοινωνία των πολιτών και ο ιδιωτικό τομέα προσανατολίζονται στο εσωτερικό εμπόριο και το ενδοκρατικό εμπόριο δηλαδή και το περιφερειακό εμπόριο. Συμφωνία GSP-SYN ε, αναφέρεται στη... στον προσανατολισμό αυτών. Αν έρθουμε τώρα στο Καμερούν. Εδώ είναι ξεκάθαρο ότι το Καμερούν πρόθεσή του δεν έχει υπογράψει ακόμα. Αλλά ο Κάρελ Ντεχούχτ έκανε μια, άκουσα μάλλον μια ανακοίνωση από την κυβέρνηση του Καμερούν που είπε ότι η πρόθεσή της είναι να υπογράψει εξαιτίας της μπανάνας. Γιατί δεν υπάρχουν δασμοί, ενώ αλλιώ θα ήταν 28%. Ενώ λοιπόν η κυβέρνηση είναι έτοιμη να υπογράψει, υπάρχουν αντιδράσεις και μέσα στην κυβέρνηση. Αλλά βέβαια οι πολιτικοί ηγέτες θα πάρουν την απόφαση στο Καμερούν. Και υπάρχει η αίσθηση στην Κεντρική Αφρική ότι η οικονομική αυτή συμφωνία εταιρική σχέση δεν είναι η λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ιδιωτικό τομέα εκεί σήμερα. Και εδώ βλέπετε τι είπε κάποια οργάνωση αγροτών που είπε ότι οι προτεραιότητες δεν είναι σαφείς. Πρέπει να έχουμε στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις εσωτερικές δομές. Να έχουμε πρόσβαση σε χρηματοδότηση, σε δάνεια κλπ. Αυτή λοιπόν είναι η γενική άποψη που επικρατεί στην Κεντρική Αφρική. Οι βουλευτές βέβαια δεν μπορούν να μιλήσουν και πολύ στο Καμερούν, αλλά κάποιοι λένε έμεσα ότι δεν θα είναι εποφελής η Συμφωνία Οικονομική Εταιρική Σχέση, αλλά είναι πάρα πολύ ευαίσθητο το θέμα αυτό στο Καμερούν. Α έρθουμε τώρα στην Κένια. Εδώ πρόκειται για τα λουλούδια, όπου απασχολούνται πάρα πολλοί άνθρωποι στον κλάδο αυτών. Υπήρξε στήριξη. Η Κένια αποτελείται από διάφορα κρατήδια. Οπότε η κεντρική κυβέρνηση πρέπει να πιστεί να υπογράψει την Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης. Και εδώ όμως, αν υπογράψει η Κένια, αυτό θα έχει επιπτώσει σε άλλους τομείς της οικονομίας. Στην Ανατολική Αφρική λοιπόν το κοινοβούλιο είναι ιδιαίτερα δραστήριο. Υπάρχει η νομοθετική συνέλευση της Ανατολικής Αφρικής και στην Κένια η κυβέρνηση είπε ότι δεν θα υπογράψει τη συμφωνία έτσι όπως έχει τώρα, εκτός αν τα θέματα των ρητρών που ζητούν, εξαγωγών λοιπά διευθετηθούν. Το θέμα των δασμών εξαγωγών επίσης είναι κάτι ενδιαφέρον. Αυτό έχει να κάνει με όλες τις πλευρές. Φαίνεται ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο το οποίο πρέπει να παραμείνει. Σύμφωνα με το Business Council της Ανατολικής Αφρικής, οι χώρες Ανατολικής Αφρικής θα πρέπει να μπορούν να επιβάλλουν δασμούς εξαγωγής για λόγους βιομηχανοποίησης. Και ε, Ας έρθουμε μάλλον τώρα στην Αμίμπια. Εδώ πέρα πρόκειται για αλλιεύματα, αλλά και για βόλιο κρέας. Έχουν πέσει πάρα πολλοί οι εξαγωγές. και οι δασμοί θα είναι ανάμεσα στο 4% και στο 19,5%. Η κατάσταση στην Αμήβια είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα για την Αμήβια. Ήδη εφαρμόζει την ε, Συμφωνία Εμπορικής Ανάπτυξης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως συμμετέχει και η Νότια Αφρική. Είναι μια συμφωνία η οποία υπογράφηκε αμέσω μετά το Απαρτχάιτ με την Νότια Αφρική και επειδή έχει τελωνιακή ένωση η Ναμίμπια με την Νότια Αφρική, έχουν δυσκολίες να συνδυάσουν ε, τις εισαγωγές από το Cape Town και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και ο Υπουργός Εμπορίου της Ναμίμπια και ο Πρωθυπουργό έχουν εκνευριστεί πολύ με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βγάλουν την Ναμίβια από τον κανονισμό 1528 του 2007. Λένε δεν μπορείτε να δράσετε μονομερός, ότι δεν είναι αυτό το πνεύμα συνεργασίας, δεν είναι αυτή η ιδέα της συνεργασίας μέσα στις συμφωνίες κανονικά. Όλα αυτά βέβαια πρέπει να τα δείτε λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ναμίμπια νιώθει ότι της γίνεται αδικία. Γι' αυτό και αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο. Αλλά υπάρχει ένα πλαίσιο βέβαια μέσα στο οποίο γίνονται λεφτά. αυτά. Μποτσουάνα τώρα. Η Μποτσουάνα εξάγει κυρίως βόηο κρέας, που επίσης θα πέσουν πολύ. Αν δεν εξάγουν βόηο κρέας, τότε δεν τους μένει τίποτα. Έχουμε μιλήσει με πολλούς παράγοντες από εκεί και λένε «Μα πρόκειται για την ανάπτυξη. Αν δεν μπορούμε να εξάγουμε βόηο κρέας, τότε ε, κάτι και δεν θα έχουν τίποτα άλλο να κάνουν». Γι' αυτό και ο υπουργό Εμπορίου είπε ότι η Μποτσουάνα ναι, να υπογράψει, να επικυρώσει. Αλλά συγχρόνως είπε ότι η Μποτσουάνα δεν έχει την επιλογή, δεν μπορεί να κάνει και τίποτα άλλο με τα Φίτζι και Σοζιλάνδη. Ζάχαρη. Στις χώρες αυτές η ζάχαρη καλλιεργείται πολύ εντατικά και απασχολούνται πάρα πολύ. Ο κλάδος για τα Φίτζι είναι αυτός που απασχολεί τον περισσότερο κόσμο. Οπότε αν χαθεί αυτό, τότε χάνεται και η οικονομία, καταστρέφεται εκεί. μου επιτρέπετε να συνεχίσω στα απορίσματα. Το κεντρικό νόημα είναι ότι η Ευρώπη, αν και το ίδιο κάνει τις τελευταία χρόνια στις διαπραγματεύσεις, τίνει να είναι πιο ε, ευέλικτη, στην ουσία δεν έχει δείξει πραγματική ευελιξία, ήταν επιφανειακή ευελιξία και τα επίμεχα θέματα στις διαπραγματεύσεις εξακολουθούν να παραμένουν χωρίς να έχει λυθεί κάποιο πρόβλημα. Για παράδειγμα, για το θέμα της εσωτερική στήριξης είναι, εξακολουθεί να είναι θέμα στις χώρες ΑΚΕ, στις περιφέρειες της Αφρικανικής κοινότητας, όπως για την πρόσβαση στην αγορά, στην περιφέρεια ΕΚΟΒΑΣ, όπως ανέφερε και ο Πίτερ, υποτίθεται ότι υπήρχε μια ευελίξια, διότι η Ευρώπη συμφώνησε στο 75%, αλλά όταν δούμε τα νούμερα και ενημερώσουμε τα στοιχεία μας, τα, τελευταία στοιχεία ανέρχεται στο 82% αν χρησιμοποιήσουμε δηλαδή πιο ενήμερα εμπορικά στοιχεία. Και για τη μεγαλύτερη οικονομία την Ιγυρία θα πρέπει να απελευθερώσουν ήδη το 81% σε 15 χρόνια και 86% σε 20 χρόνια. Για το θέμα των ε, εξαγωγικών δασμών που είναι ιδιαίτερα επίμαχο σε πολλές υποπεριφέρειες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον ε, το Ανατολικό Αφρικανικό Συμβούλιο έχει διαπραγματευτεί τη δυνατότητα εισαγωγής νέων εξαγωγικών δασμών, αν αυτό είναι απαραίτητο, αλλά τώρα το λένε αυτό μόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο για μια περιορισμένη χρονική διάρκεια και μόνο με την ε, έγκριση του Συμβουλίου ε, της ε, εταιρικής σχέσης που συμπεριλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως. Εξαρτάται δηλαδή από τους υπουργούς και μένει εκρεμές το θέμα. Πώς λοιπόν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Έχουμε την εντύπωση ότι οι τεχνικές συζητήσεις μπορούν να συνεχίζονται επάπειρον, αλλά δεν θα λύσουν κάποιο πρόβλημα. Βεβαίως μπορεί να επικρατήσουν τρία διαφορετικά σενάρια. Το ένα είναι ότι οι ευρωπαϊκές χώρες μπορεί να αρνηθούν να συμβιβαστούν λόγω αυτών των πιο μακροπρόθεσμων στόχων επιθυμούν βιομηχανοποίηση και άρα χρειάζονται τους δασμούς για να στηρίξουν τη διαδικασία βιομηχανοποίησης ή μπορεί και να καταρρεύσουν υπό την πίεση, διότι χρειάζονται και επιθυμούν αυτή την προτιμησιακή πρόσβαση. Τρίτο σενάριο, δυνητικό σενάριο, είναι κάποιος να αρνηθεί, κάποιες χώρες να αρνηθούν την συμφωνία, ενώ άλλες να τη δεχτούν, όπου βεβαίως θα επικρατεί σύγχυση. Ούτω ή άλλως θα έχουμε ε, ε, την απειλή, απειλές για την περιφερειακή ολοκλήρωση, γιατί το εμπόριο είναι διαφορετικό στις διάφορες περιφέρειες ή γιατί το περιφερειακό εμπόριο, ακόμα και αν όλοι δεχτούν την ε, συμφωνία εταιρική σχέσης και έχουμε ένα κοινό εμπορικό καθεστώς, πιθανότητες είναι ε, ότι οι χώρες αυτές θα πλημμυρίσουν από ευρωπαϊκά προϊόντα και όχι από περιφερειακά. Αυτό θα έχει αντίκτυπο στο περιφερειακό εμπόριο και στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η Ευρώπη λοιπόν έχει δύο τρόπους που μπορεί να αντιδράσει. Όπως προκύπτει από τους διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς με τους καταρχήν να παρουσιάσει επιλογές όπως ε, οι γενικευμένες προτιμήσεις ε, ΣΥΝ, μεταρρύθμιση των γενικευμένων προτιμήσεων, εξαίρεση για την Αφρική, ώστε να, όπως ας πούμε το, ο νόμος για την ευκαιρία ανάπτυξη στην Αφρική, όπως έχουν οι ΙΠΑ. Ε, και το 2011 η Αφρικανική Ένωση υπέβαλε πρόταση για τις προτιμήσεις όπου βασικά αναφέρει πως ε, η ε, Τελωνιακή Ένωση των λιγότερων ανεπτυγμένων χωρών θα πρέπει να τυχαίνει τις ίδιες μεταχείρισης όπως και οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, δηλαδή ε, όλα εκτός από όπλα. Και αυτή είναι η πρότασή τους, ώστε να υπάρξει μια μικρή βελτίωση του προγράμματος γενικευμένων προτιμήσεων ε, για τις ε, λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και τους γειτονές τους. Συγγνώμη, πρέπει να τελειώνετε. Έχετε ξεπεράσει το χρόνο σας εδώ και τρία λεπτά. Ναι, κλείνω. Να έχουμε δηλαδή ένα είδος ε, πίνακα επιδόσεων ώστε να βλέπουμε ποιο είναι το επίπεδο απελευθέρωσης ε, ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης της κάθε χώρας και δεύτερον Ίσως ε, το πρόγραμμα GSP συν να γίνει πιο ευέλικτο. Τρίτον, να μεταρρυθμιστεί το σύστημα GSP για να ληφθούν υπόψη τα όσα έχουν συμφωνήσει το 2011 οι Αφρικανοί Υπουργοί Εμπορίου. Και τέταρτον, μια εξαίρεση για την Αφρική όπως έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Μολδαβία, τα Δυτικά Βαλκάνια και για το Πακιστάν. Δεν έχουμε χρόνο, αλλά αυτή είναι η λογική που έδωσε η Ευρώπη. Ε, ναι, όχι, δεν έχετε άλλο χρόνο, διακόπτη πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ. This is a very important question. Πολύ σημαντικό θέμα. Σας ευχαριστώ για την εισήγησή σας. Περιγράφεται μια κατάσταση που είναι φρικτή για το Καμερούν την Ναμίβια, την Κένια, την Μποτζουάνα, την Ιγυρία. Like to uh, hear questions from... Και τώρα θα ήθελα να ακούσω ερωτήσεις από τα μέλη αν υπάρχουν και τη γνώμη της Επιτροπής για αυτή την κατάσταση. Yes. No, nobody wants. Yes. So, um, I should like to... Λοιπόν, Να ακούσουμε τον κύριο Βάλα για την κατάσταση αυτή που έχει δημιουργηθεί. Όπου ασκείται πίεση και καταστρέφεται η αγορά σε αυτές τις χώρες. Well, thank you for the... Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για αυτή την εισήγηση. Τα τελευταία χρόνια σε αυτή την Επιτροπή παρακολουθείτε πάντοτε από κοντά της ε, ΕΠΑ και εκτιμούμε τις ευκαιρίες που μας δίνετε να απαντήσουμε στις ε, ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ που μας προσκαλέσατε. Θέλω να ευχαριστήσω και τους εισηγητές αυτής της μελέτης. Για αυτή τη μελέτη που είναι μια συλλογή ε, θέσεων σχετικά με τις ΕΠΑ, τις οποίες ήδη γνωρίζαμε και στις οποίες θα επανέλθουμε εντός ολίγου. Πρόεδρε, νομίζω πως είναι σημαντικό να, κάνουμε, να πούμε τα εξή. Να πω τα εξή στο χρόνο που μου διαθέτετε. Το πρώτο είναι ότι είπα δεν προέκυψαν εκ του μηδενός, είναι κοινέ ε, ε, συμφωνίες που προκύπτουν από τη Συμφωνία του Κοτονού. Στόχο είχαν τρία πράγματα. Πρώτον, να αντικαταστήσουν τις μονομερείς εμπορικές προτιμήσεις από κάτι πιο ισχυρό, να παρέχουν προβλεψιμότητα και σταθερότητα σε εμπορικές σχέσεις ε, ε, και συμμόρφωση προς τον ΠΟΕ, καθώς και να εισάγει την ε, απελευθέρωση του εμπορίου ώστε να προωθηθούν οι επενδύσεις, η ανταγωνιστικότητα και να χρησιμοποιηθούν ως ένα εργαλείο για την ανάπτυξη. Εάν επανέλθουμε λοιπόν σε αυτή την κοινή, στο κοινό όραμα και δούμε ότι οι εναλλακτικέ που προσφέρθηκαν δεν κάνουν κανένα ή μπας περιπτώσει όλα από αυτά τα πράγματα, Επίσης το ότι το ΕΠΑ ε, στην ουσία κινούνται πολύ αργά. Είδαμε ότι τρεις ΕΠΑ πέρασαν στη φάση της εφαρμογής. Είδαμε την έγκριση διαφόρων συμφωνιών από το Κοινοβούλιο, πάλι για τον Ειρηνικό. Κεντρική Αφρική, Καμερούν και ο, η τροποποίηση του κανονισμού για την πρόσβαση στην αγορά υπερψηφίστηκε από συντριπτική πλειοψηφία εδώ στο Κοινοβούλιο. Κάνουμε πράγματα δηλαδή από κοινού, ξεκινάει η εφαρμογή και το πιο σημαντικό είναι ότι οι διαπραγματεύσεις πετυχαίνουν αποτελέσματα. Παρά τις ε, ε, τα παράπονα για έλλειψη ευελιξίας. Έχουμε αποτελεσματικά καλύψει το κενό με την Δυτική Αφρική και υπάρχει και ένα σχέδιο συμφωνίας που εγκρίθηκε από τους επικεφαλείς των διαπραγματεύσεων και τώρα περιμένουν για, περιμένει για την πολιτική του έγκριση. Επίσης έχουμε λύσει πολλά θέματα με και μέσα στην δυτική, δυτικοαφρικανική κοινότητα μέσω αυτών των διαπραγματεύσεων. Οπότε πιστεύω, Πρόεδρε, πως δεν μπορούμε να μιλάμε για τις ΕΠΑ χωρίς να αναφέρουμε και αυτό το κομμάτι της εικόνας, το θετικό. Και αυτό είναι και κάτι που με στενοχωρεί για την σημερινή συζήτηση ότι εξετάζει τις απειλές που απορρέουν από τη ΕΠΑ με την προϋπόθεση ότι η απελευθέρωση του εμπορίου είναι αρνητική και ίσως και βλαβερή, ενώ δεν μιλά για αυτό το κοινό όραμα που είχαμε για μια ΕΠΑ που θα αυξάνε ε, τις επενδύσεις ε, και την ανάπτυξη και θα ε, έφερνε επενδύσεις. Και όλες οι ευελιξίες που δόθηκαν και που είναι πολύ γνωστές σε όσους παρακολούθησαν τις διαπραγματεύσεις θα πρέπει και αυτές να αναφέρονται διότι οι εξαιρεσει που δεχτήκαμε επιτρέπουν στους εταίρους μας να εξαιρούν όλα τα ευαίσθητα προϊόντα, ενώ υπάρχουν και ασφαλιστικά μέτρα που καθυστερούν την απελευθέρωση και τους επιτρέπουν να αντιμετωπίσουν και άλλες προκλήσεις συμπεριλαμβανομένων των εσόδων. Το έγγραφο το οποίο η μελέτη που μας παρουσιάστηκε σήμερα, ενώ είναι μια καλή συλλογή διαφόρων απόψεων σε σχέση με τις ΕΠΑ, δεν παρέχει κριτική ανάλυση αυτών των δηλώσεων και δεν γίνεται καμιά απόπειρα για ε, εξισορρόπηση με τις πιο θετικές δηλώσεις που και εμείς έχουμε ακούσει στη διάρκεια των ετών. Οπότε, νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε να δούμε ε, την ε, κοινέ αυτέ εταιρικέ σχέσει, τι οποίε έχουμε προβεί, να αναγνωρίσουμε ότι έχει σημειωθεί πρόοδο στι διαπραγματεύσει και να στηρίξουμε με όλη μα την ενέργεια την επιτυχία τη εφαρμογή αυτών των συμφωνιών. Σα ευχαριστώ που μου δώσατε το χρόνο να το εξηγήσω αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Άσκολα. Ή η κυρία Άσκολα. Διορθώνει πρόεδρος. ο προεδρος επιθυμειτε το λόγο? Όχι. Καλώς. Θα δώσω τότε το λόγο και πάλι στους δύο συντάκτες της μελέτης για πέντε λεπτά παρακαλώ για να ολοκληρώσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να απαντήσω λέγοντας πως όσον αφορά την ε, συμφωνία του Κοτονού υπήρχε το άρθρο 37 που κατά βάση έλεγε πως όταν τα συμβαλόμενα μέρη δεν θεωρούν πως είναι σε θέση να υπογράψουν τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης, θα πρέπει να έχουν κάποιες εναλλακτικέ λύσεις που θα τους δίνουν εξίσου καλές προτιμήσεις. Όσον αφορά το ζήτημα της απελευθέρωσης του εμπορίου και το υπόδειγμα που αντικαθιστά το μοντέλο προτιμησιακής μεταχείρισης ήταν πολύ ενδιαφέρον γιατί η Ευρώπη όταν απίθυνε έκκληση ε, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου για μη αμοιβαία προτιμησιακή μεταχείριση των Δυτικών Βαλκανίων είπε πως το να τερματιστούν οι προτιμήσεις θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στα Δυτικά Βαλκάνια και έτσι στις ε, διαδικασίες ε, μεταρρυθμίσεων επιπλέον δεδομένης της Παγκόσμια οικονομικής επιβράδυνσης θα μπορούσε να κινδυνεύσει η οικονομία των χωρών αυτών. Όταν έκανε μια ανάλογη έκκληση για την Μολδαβία η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε πως η Μολδαβία είναι η φτωχότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Υπήρου και ήταν αναγκαίο να προσφερθεί στη Μολδαβία βελτιωμένη πρόσβαση στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αναπτυχθεί η οικονομία της μέσω αυξημένων εξαγωγών. Γιατί λοιπόν αν λειτουργεί τόσο, καλά, Εάν δεν λειτουργεί τόσο καλά στη Μολδαβία και τη Δυτική Αφρική, γιατί να λειτουργεί τόσο καλά στην Αφρική. Για το θέμα της έκοβας ε, της κοινότητας αυτής, ναι υπήρχε ένα σχέδιο συμφωνίας στο επίπεδο εμπειρογνωμόνων, αλλά τώρα πρέπει να επανέλθει στις χώρες και να ληφθεί μια αποφασία από τους υπουργούς, ε, τους αρχηγούς κρατών μελών και αυτό το οποίο ακούσαμε ήταν πως οι Νιγηριανοί οργάνωσαν ένα εργαστήριο σχετικό ενδιαφερομένων και από ό,τι φαίνεται η Νιγηρία θα απέριπτε την συμφωνία γιατί θεωρούσαν πως θα ήταν συνέπειες για την εσωτερική οικονομία και ο κύριος Υπουργό απέθυνε μια επιστολή στον πρόεδρο της Νιγηρίας για να εξηγήσει την κατάσταση και να ζητήσει από τον πρόεδρο να λάβει μια απόφαση. Οπότε δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική απόφαση αλλά νομίζω πως οι ενδιαφερόμενοι στην Νιγηρία αποφάσισαν έτσι. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει η Έκοβάση κοινότητα αυτή. Απλά θα ήθελα να πω πως ε, τα ζητήματα αυτά ε, παραμένουν στις διάφορες ε, περιφέρειες. Just for me to thank... Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω. Θεωρώ πως η Επιτροπή μας ε, θα παρακολουθήσει οπωσδήποτε αυτό το ζήτημα και στην επόμενη θητεία. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης πλατφόρμα για τον συνδυασμό μέσω στην εξωτερική συνεργασία. Εδώ πρόκειται για μια ενημέρωση όσον αφορά τις συνεδριάσεις αυτής της πλατφόρμας εν ώψη της επόμενης συνεδρίασης της ομάδας πολιτικής που θα γίνει στις 4 Απριλίου. Όπως γνωρίζετε στις 27 Απριλίου στείλαμε μια επιστολή στον Επίτροπο Πίπαλξη και στην Βαρόνη Άστον για να υπογραμμίσουμε τις ανησυχίες μας σε σχέση με διάφορες πτυχές της μεταρρύθμισης των διατάξεων όσον αφορά το συνδυασμό μέσων. Blending facilities στα αγγλικά. Ο κ. Μπάκσταρς έπρεπε να σας παρουσιάσει τα πρακτικά αυτής της διαδικασίας, όμως ο κύριος Στάς δεν μπόρεσε να είναι σήμερα εδώ και μου άφησε το σημείωμα για την εισήγησή του, οπότε θα σας το διαβάσω. Οπότε θα το διαβάσω εξ ονόματός του. je στα αγγλικά είναι το σημείο μου, οπότε θα αλλάξω γλώσσα. Όπως ξέρετε, το Δεκέμβριο του 2012 η πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον συνδυασμό μέσων στην εξωτερική συνεργασία επεκτάθηκε. Η πλατφόρμα αυτή βεβαίως είναι υπό την ηγεσία μιας ε, ομάδας ε, πολιτικής και έχει τη στήριξη τεχνικών ομάδων. Ο συσυγητής, ο κύριος Στάς, παρακολουθεί στενά τη δουλειά της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας και θα ήθελε να συζητήσει μαζί σας κάποια βασικά ζητήματα τα οποία επίσης θα είναι στην μερίσια διάταξη που βεβαίως ε, προγραμματίζεται για τις 4 Απριλίου. Όπως είπαμε, τον Ιανουάριο απευθύναμε μια επιστολή στον ε, Επίτροπο Πίμπαλξ και την κυρία Άστον και παρουσιάσαμε τις ανησυχίες μας. Η απάντηση της Παρασκευής ε, έδωσε κάποια διαβεβαίωση, αλλά βεβαίως σεβασμός τον βασικών στόχων της δημοκρατικής ε, δομής και της διοίκησης, η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι πολύ σημαντικά ζητήματα. Όπως γνωρίζετε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφέρει πως από την σκοπιά της ανάπτυξης το νέο αυτό μέσο δεν θα πρέπει να έχει άλλο σκόπο πέραν από τη μείωση της φτώχειας και την καταπολέμηση της ανισότητας και ζητάει από την ευρωπαϊκή κοινότητα να δώσει σαφείς πληροφορίες για το πώς ο μηχανισμός αυτός εξυπηρετεί το σκοπό μιας αναπτυξιακής πολιτικής που βασίζεται στα κριτήρια αυτά και στο πώς οι δυνατότητες του Κοινοβουλίου θα μπορέσουν να ασχηθούν. Επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επεσήμανε στις προπαρασκευαστικές συναντήσεις ε, του στρατηγικού διαλόγου πως θα πρέπει να υπάρξει μία ανάπτυξη η οποία δεν θα μειώσει καθόλου τη φτώχεια. Επίσης παρατηρούμε πως κατά βάση αυτή τη στιγμή εστιάζουμε σε επενδύσεις σε υποδομές μεγάλης κλίμακας με στόχο να προχωρήσουμε σε κάποια περαιτέρω ανάπτυξη που υποτίθεται πως θα βοηθήσουν έτσι την γενικότερη ανάπτυξη. Επίσης, βλέπουμε πως αυτό προβλέπεται και για νέους τομείς όπως η εκπαίδευση, η ανάπτυξη της υπαίθρου και διάφορα γεωγραφικά προγράμματα, οπότε δεν αφορά μόνο μεγάλα ενεργειακά έργα. Δεδομένου του ότι ο ιδιωτικός τομέας θα επενδύσει μόνο εάν μπορεί να υποφεληθεί από κάτι, νομίζω πως πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί εάν ε, το χρησιμοποιούμε αυτό μόνο για τους κοινωνικούς τομείς ή την ανάπτυξη της υπαίθρου. Θα ήθελα τώρα να θέσω τα εξής ερωτήματα. Πώς μπορεί να συνεισφέρει αυτό. Πώ μπορεί να συνεισφέρει αυτό που συμφωνεί στη μέση της φτώχειας στις ε, αγροτικές περιοχές, να βοηθήσει την αηφόρο χρήση ενέργειας από μικρές από ε, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πώς μπορεί η Κομισιόν να διασφαλίσει πως δεν θα οδηγήσει ανταυτού στην επέκταση της μόνο καλλιέργειας που δεν ανταποκρίνεται στις τοπικές ανάγκες αλλά στις μεγάλες επιχειρήσεις. Επίσης, πώς μπορεί η δυνατότητα αυτή να απαντήσει στους ε, στις ανάγκες των ευπαθών ομάδων. Δεν είναι γεγονός ε, πως ε, θα διηγηθούμε έτσι σε ένα σύστημα δύο ταχυτήτων με πλήρη αντίφαση στο ζήτημα της ε, εκπαίδευσης και πώς θα διασφαλίσουμε ότι οι ε, δυνατότητες αυτές ε, θα βοηθήσουν την ικανότητα μόχλευσης των επενδύσεων για, το, για περιοχές στις οποίες μπορεί κανείς να έχει δύσκολα πρόσβαση χρηματοδοτούντας παραδείγματος χάρη πρωτοβουλίες ανάπτυξης των φτωχών ή που θα έχουν απόδοση υψηλότερη από τον χρηματοοικονομικό ειδικά όταν υπάρχουν ιδιώτες. Πώς θα δοθεί κίνητρο για τέτοιες επενδύσεις, ποια είναι τα κατάλληλα μέσα, για ποιον κλάδο. Αυτό δεν είναι ακόμα ε, σαφές. Αναμένουμε από την Κομισιόν και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να δώσουν σαφείς οδηγίες αντιπροσωπείες για να επιτύχουμε αυτούς τους σημαντικούς στόχους. Συγκεκριμένα πρέπει να υπάρξουν διασφαλίσεις για το ότι η χρήση ε, αυτή δεν θα οδηγήσει σε αύξηση τελών χρηστών βασικών υπηρεσιών. Όσον αφορά το στόχο μείωσης της στόχιας, καλωσορίζουμε το ότι οι μελλοντικές αιτήσει θα συμπεριληφθούν και ακόμα θεωρούμε πως η αξιολόγηση ex ante απαιτείται για κάθε έργο όπως προτείνεται στην μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όσον αφορά την διαχείριση του μηχανισμού συνδυασμού. Πρέπει να δούμε τη δημοκρατική διάσταση. Καλωσορίζουμε το ότι η Κομισιόν και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης καλωσορίζουν την διαδικασία αυτή ευθύς εξ αρχής. Όπως ήδη είπαμε στην επιστολή μας θεωρούμε πως για να διασφαλιστεί αποτελεσματική ε, αυτή αρχή θα πρέπει να συνδυάσουμε και την στρατηγική και την επιχειρησιακή πτυχή. Θα μπορούσε η Κομισιόν και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να ε, επεκταθεί σε αυτό το θέμα, ειδικά όσον αφορά την ε, την συμμετοχή των χωρών αυτών στην στρατηγική και την στρατηγική και την επιχειρησιακή. Πρόσφατες μελέτες ε, για το μέσο αυτό η Κομισιόν και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης έχουν διασφαλίσει πως το στοιχείο αυτό της τεχνικής αρρωγής συχνά συμπεριλαμβάνεται σε ένα επενδυτικό έργο. Εμεί θεωρούμε το, στο ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ελπίζουμε πως στο μέλλον η Κομισιόν και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα κατανείμουν τους πόρους αυτούς για να χρηματοδοτηθεί η δυνατότητα αυτή η απόκτηση ικανοτήτων. Επίσης υπάρχει και ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών και η παρακολούθηση και αξιολόγηση του αντικτύπου των έργων που χρηματοδοτούνται. Η Κομισιόν ήδη έχει δοκιμάσει το μοντέλο αυτό με τις οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών όσον αφορά την στήριξη από τον προπολογισμό. ζητήσαμε ο ενδιαφερό, οι ενδιαφερόμενοι πληθυσμοί να συμμετέχουν σε όλες τις διαδικασίες ε, του συνδυασμού μέσων θεωρούμε πως θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος της τοπικής κοινωνίας των πολιτών κατά τη φάση της εφαρμογής ενισχύοντας τον ρόλο τους. Θα μπορούσε η Κομισιόν και η Υπηρεσία εξωτερική δράση να επεκταθούν στο ζήτημα αυτό ξεκαθαρίζοντας το πώς σκοπεύουν να συμπεριλάβουν ενεργά τις οργανώσεις της κοινωνία των πολιτών, της κοινωνίας των πολιτών αναγνωρίζοντας τον ρόλο τους. Όσον αφορά δε την συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας των Πολιτών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε όχι μόνο ενημέρωση αλλά και εμπλοκή στην συζήτηση της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας ε, για το Συνδυασμό Μέσων. Θα μπορούσε η Κομισιόν και η Υπηρεσία Εξωτερική Δράση να εξετάσουν την δυνατότητα πρόσκληση τη κοινωνία των πολιτών σε μελλοντικέ τεχνικέ συναντήσει τη πλατφόρμα για να υπάρχει αποτελεσματική συμμετοχή του. Τέλο, όσον αφορά το ζήτημα της διαφάνειας ε, και της λήψης αποφάσεων. Θα ήθελα να υπενθυμίσω κάποια ζητήματα. Τα κριτήρια επιλογής έργων πρέπει να δημοσιοποιηθούν ε, και έτσι να δοθούν πληροφορίες ε, εγκαίρως. Ε, χρειάζονται επίσης περισσότερες διευκρινήσεις στο ζήτημα της διαφάνειας και της λογοδοσίας. θεωρώ πως ο περιορισμός του κινδύνου και η χρήση τέτοιων μέσων όπως εγγυήσεις θα πρέπει να αξιολογηθούν προσεκτικά πριν ε, θεωρούμε πως ε, είναι κάποια εξωτερική βοήθεια. Τέλος, η τελευταία παρατήρηση αφορά την διαδικασία έγκρισης της ε, του συνδυασμού μέσων, κάτι το οποίο στο μέλλον δεν θα συμπεριλαμβάνει τις λεπτομέρειες του ενδιαφερόμενου φορέα. Κομισιόν και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης λένε πως αυτή τη στιγμή εγκριθούν τα έργα θα υπάρξει μια ad hoc απόφαση της Κομισιόν για να δοθούν πληροφορίες για τον ενδιαφερόμενο φορέα. Μετά την έγκριση του δημοσιονομικού κανονισμού θεωρούμε πως η απόφαση αυτή για την κάθε επιχειρήση θα πρέπει να λαμβάνεται ε, με βάση την ε, κανονική διαδικασία επιτροπολογίας κάτι το οποίο σημαίνει καλύτερη εμπλοκή των θεσμικών οργάνων, των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δίδοντας έτσι μεγαλύτερη νόμιμοποίηση και ενισχύοντας την διαφάνεια της ε, διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Θα μπορούσατε να διευκρινίσετε ποιοι είναι οι βασικοί περιορισμοί ε, για να μπει ε, εδώ πέρα η βασική διαδικασία επιτροπολογίας. Θεωρώ πως εάν έχουμε κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες δεν θα συμπεριλαμβάνονται στο ετήσιο σχέδιο δράσης ε, οι δυνατότητες του Κοινοβουλίου για κοινοβουλευτικό έλεγχο δεν θα ασκηθούν πλήρως. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω την άποψή σας επί των ζητημάτων αυτών. Σας ευχαριστώ. So, are there some... Υπάρχουν σχόλια παρακαλώ σε σχέση με τα όσα αναφέρει ο Μπαρτστάς. Τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. για αυτό το θέμα έχουμε τον κύριο Ρέις Κοντέ. Ευχαριστώ. Έχω πέντε λεπτά. Σωστά. Όσοι ήθιστε. Για να ξέρω. Πέντε λεπτά μου δίνετε. Σωστά, πέντε λεπτά έχω. Ναι, ναι, μετά από όλα αυτά που είπα εγώ, εσείς ταξίσατε και 15 λεπτά. Καλώς, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Για μας, το σημείωμα του κύριου Στάις που απευθύνει στην κυρία Στον και τον κύριο Πίλμπαξ από πλευράς της Επιτροπής αξίζει κάθε προσοχή. Και εμείς, και κύριος Στάες το λέει, ότι στα κύρια ζητήματα έχουμε ήδη απαντήσει. Είναι προφανές ότι για μας, στα πλαίσια του blending, της μίξης αυτής κονδυλίων, δεν μπορούμε να φανταστούμε προγράμματα για τα οποία οι χώρες παίρνουν δάνεια, αν οι χώρες εταίροι δεν συμφωνούν με τα προγράμματα αυτά. Η συμμετοχή δηλαδή των χωρών εταίρων είναι κεντρική σημασίας στην χρηματοδότηση των προγραμμάτων μέσω του blending. Άρα η συμμετοχή των χωρών εταίρων πρέπει να γίνεται και σε επίπεδο συζητήσεων για τον προσανατολισμό των διευκολύνσεων, των μέσων, αλλά κατά τη γνώμη μας και απευθείας σε σχέση με το κάθε πρόγραμμα, γιατί δεν είναι δυνατόν, είναι αδιανόητο να υπογράφεται από τις χώρες δικαιούχους κάποια συμφωνία χρηματοδότησης αν δεν συμφωνούν με το πρόγραμμα. Συγγνώμη, έχω μπερδέψει λίγο εδώ τα χαρτιά μου. Α, να τα βρήκα. Λοιπόν, θέλω να διευκρινίσω ένα βασικό σημείο εδώ. Στα πλαίσια του blending, 95% των δράσεών μας μέχρι τώρα, και δεν νομίζω ότι αυτό θα αλλάξει δραστικά, τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον, τα περισσότερα προγράμματά μας χρηματοδοτούνται όχι τόσο από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά από το δημόσιο. Δηλαδή, τα προγράμματά μας, όπου στο MR8 έχουμε χρηματοδοτήσει με blending προγράμματα στα πλαίσια των δημοσιονομικών προτικών των προηγούμενων 7 ετών, Είχαμε βέβαια κάποια προγράμματα για τα οποία στηριχθήκαμε στον ιδιωτικό τομέα, αλλά το 90-95% δεν ξέρω να σας πω ακριβώς, αλλά μπορώ να σας το πω αργότερα με η χρηματοδότηση έχει γίνει από το δημόσιο με δάνεια και η συμμετοχή της Επιτροπής μέσω επιδότησης επιτρέπει στις χώρες αυτές να μειώσουν τα δάνειά τους και να πετύχουν πρώτα απ' όλα να πετύχουν ρήτρε παραχώρησης ή τα δάνειά τους να τα πάρουν με τέτοιο κόστος, ώστε με κάποια επιπλέον μέσα να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν μεγαλύτερα προγράμματα από ό,τι θα είχαν χρηματοδοτήσει αν είχαν μόνο τα κοινοτικά κονδύλια ή άλλα. Και είναι σημαντικό αυτό, διότι όσα αναφέρονται στην επιστολή του κύριου Στάες για τον ρόλο του ιδιωτικού τομέα, είναι προφανές ο ότι εφόσον χρηματοδοτούμε μέσω του ιδιωτικού τομέα κάποια προγράμματα, σε συνδυασμό βέβαια με κρατικές τράπεζες, γιατί πάντα συνεργαζόμαστε διμερός. Είναι προφανές λοιπόν ότι πρέπει να διασφαλίσουμε πως η συνεισφορά των τραπεζών, δημοσίων και ιδιωτικών, δεν υπερβαίνει και δεν ε, είναι πέρα από τους στόχους ανάπτυξης, γιατί οι στόχοι ανάπτυξης είναι αυτοί που καθορίζονται για τη συνεργασία μας. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν πρέπει να δούμε την χρηματοδότηση μέσω της μίξης κονδυλίων, μέσω του blending για υποδομές, κοινωνικές υπηρεσίες, εκπαίδευση. Ό,τι έχει γίνει κατά το παρελθόν η χρηματοδότηση η ιδιωτική στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης είναι κάτι που πρέπει να δούμε λαμβάνοντας υπόψη τη χρηματοδότηση του δημοσίου τομέα που οδηγεί στη δυνατότητα δάνειοδότησης για την χρηματοδότηση της εκπαίδευσης και της υγείας που αλλιώς δεν θα ήταν εφικτή. Αυτή είναι η οπτική γωνία από την οποία πρέπει να εξετάζουμε το θέμα της χρηματοδότησης, της υγείας, της εκπαίδευσης και άλλων κοινωνικών τομέων. Το blending δηλαδή πρέπει να χρησιμοποιείται, και αυτό έχει γίνει μέχρι τώρα και πρέπει να συνεχιστεί, πρέπει να χρησιμοποιείται για να μπορούμε να ενισχύσουμε επιπλέον δημόσιες επενδύσεις, οι οποίες δεν θα είχαν λάβει χώρα εάν δεν υπήρξε η δικιά μας η αρρωγή. Γιατί δεν θα μπορούσαν να είχαν πετύχει δάνεια σε τιμή αποδεκτή για τις χώρες αυτές. Εδώ έρχομαι και στο θέμα της συμμετοχής των χωρών εταίρων και στο ρόλο των χωρών αυτών στη διακυβέρνηση. Παρακολουθήσαμε προσεκτικά τις συστάσεις, τις συμβουλές, τις προπτικές που έδωσαν οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ομάδα της πλατφόρμας. Είναι σαφές ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφισημία. Οι χώρες δικαιούχοι, οι χώρες εταίροι πρέπει να παίζουν σημαντικό ρόλο σε κάθε δράση. Και αυτό μόφανα δεν είναι μόνο από την πλευρά της Κομισιόν, το είδαμε αυτό στην πλατφόρμα και από τις χώρες μέλη και από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ο διάβολος βέβαια βρίσκεται στη λεπτομέρεια όπως λέμε. Πώς δηλαδή να διασφαλίσουμε τη συμμετοχή αυτή των χωρών δικαιούχων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι προφανές ότι χρειάζεται συζήτηση επί της στρατηγικής με τις χώρες εταίρους, συζήτηση για τις κατευθυντήριες γραμμές, για το pipeline. Είναι συζήτηση που πρέπει να γίνεται απευθεία με τις χώρες εταίρους. Κατά τη γνώμη μας όμως, θα είναι πολύ καλύτερα αν αυτό γίνεται στις υπάρχουσες δομές και όχι να δημιουργήσουμε ad hoc δομές όπως έγινε κατά το παρελθόν με τα Boss Strategic και είναι καλύτερα να βρισκόμαστε σε ήδη υπάρχουσες δομές. Τουλάχιστον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό πιστεύει. Πρότασή μας λοιπόν για το blending και την διαχείριση της διευκόλυνσης είναι να μην καταργηθεί η συζήτηση, αλλά η συζήτηση αυτής στρατηγικής σημασίας να γίνεται στα πλαίσια ήδη υπαρχουσών δομών και όχι να δημιουργούμε νέες δομές. Παίρνουμε μεγάλη σημασία στη συζήτηση αυτή. Στην περίπτωση, μάλιστα, που οι δομές αυτές δεν υπάρχουν, πρέπει να δημιουργηθούν. Πρέπει να υπάρχει δηλαδή αυτό το board, ε, strategic board, έτσι ώστε να γίνεται η συζήτηση. Κάτι άλλο σημαντικό είναι ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών. Πιστεύουμε ότι έχουμε όλες συμφέρον για να στηρίξουμε τα προγράμματα μέσω του blending, να έχουμε την άποψη και των τοπικών αρχών αλλά και της κοινωνίας των πολιτών για προγράμματα τα οποία έτσι και αλλιώς χρεώνουν τις χώρες εταίρους. Είναι προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από κοινού. Συνεπώς, πρέπει να γίνεται συζήτηση και με την κοινωνία των πολιτών και με τις αρχές και την κοινωνία των πολιτών. Είναι κάτι ιδιαίτερα θετικό για την ποιότητα τελικά των προγραμμάτων. Γι' αυτό και πιστεύουμε ότι οι αντιπροσωπείες μας είναι οι καλύτερες, στην καλύτερη θέση προκειμένου να βοηθήσουν στη συζήτηση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη την επιθυμία όλων των πλευρών στο σχεδιασμό, τη σύλληψη αλλά και την ε, εκτέλεση των ε, προγραμμάτων. Πιστεύουμε ότι πρέπει να ενισχυθεί λοιπόν ο ρόλος των αντιπροσωπιών μας, να ενισχυθεί ο ρόλος των αντιπροσωπιών μας στα πλαίσια της παρουσίασης του έργου πρώτα απ' όλα. Και στη συνέχεια να ενισχύεται ο διάλογος με τις χώρες εταίρους, τις τοπικές αρχές, την κοινωνία των πολιτών για να ενισχυθεί η διαφάνεια γύρω από κάθε πρόγραμμα που χρηματοδοτούμε. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι πρόβλημα περισσότερη διαφάνεια στο blending. Θέλουμε να είναι πιο ξεκάθαρη η κατάσταση και είναι μια προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε και στην τεκμηρίωση που έχουμε για τον προγραμματισμό, για την επιλογή των προγραμμάτων, για τον εντοπισμό των τομέων. Γιατί είναι σαφές ότι το blending δεν είναι η απάντηση σε όλα τα προβλήματα χρηματοδότησης που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη. Το blending είναι ένα μέσο, ένα εργαλείο που πρέπει να χρησιμοποιείται στις κατάλληλες συνθήκες και με τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Άρα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στα κριτήρια τα οποία μας οδηγούν να αποφασίζουμε για blending σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και να είναι σαφές γιατί επιλέγεται το ένα ή το άλλο πρόγραμμα. Θα υπάρξει συνάντηση της πλατφόρμας στις 4 Απριλίου με συμμετοχή των χωρών μελών. Ελπίζουμε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκπροσωπηθεί εκεί. Οι παρεμβάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις συνεδριάσεις αυτές είναι πολύ σημαντικές κατά την άποψη της Κομισιόν, γιατί δείχνουν τη βούληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συμμετέχει στη συζήτηση αυτή για το blending. Άρα πολιτικά έτσι ενισχύεται η ατζέντα. Στις 4 Απριλίου νομίζω ότι θα έχουμε ένα σχεδιασμό για την μελλοντική διαχείριση της διευκόλυνσης αυτής και θα συζητήσουμε για μελλοντικό πρόγραμμα δράσης και θα έχουμε ένα σαφή σχεδιασμό του τι είναι η διαχείριση της διευκόλυνσης αυτής. Επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια και για την επιτροπολογία. Αυτό το οποίο προτείνεται στο governance document, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση με το Κοινοβούλιο και τις κυβερνήσεις, αυτό που προτείνεται είναι αυτό ακριβώ που κάνουμε και τώρα. Δεν προτείνεται τίποτα το οποίο μειώνει το βαθμό ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή τη συμμετοχή των κρατών μελών. Αυτό που καλούμεθα να κάνουμε εξαιτία του Μοσιονομικού κανονισμού βάσει της απόφασης της Επιτροπής για να αποφασίζει για το ένα ή το άλλο πρόγραμμα, προσθέτουμε ένα επιπλέον στάδιο. Δεν προτείνουμε καμία μείωση σε σχέση με το τι κάνουμε σήμερα. Δεν βγάζουμε τίποτα. Αντίθετα, περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται στα πλαίσια των ΑΠΕ. Θα υπάρχουν και περισσότερα στοιχεία στο reporting. Υπάρχει επίσης η υποχρέωση που τα προβλέπει αυτά δηλαδή ο δημοσιονομικός κανονισμός. Δεν μειώνεται σε τίποτα ο έλεγχος ή η ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αντίθετα. Προστίθεται ένα επιπλέον τεχνικό στάδιο. Αλλά για τα θέματα αυτά της επιτροπολογίας, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να μας δοθεί ευκαιρία να συζητήσουμε περισσότερο, να δοθούν περισσότερες διευκρινήσεις από εμά ή αν είναι εντελώ ξεκάθαρο αυτό το ζήτημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ για τα σχόλια αυτά. Μας λέτε λοιπόν ότι 1,8 δισεκατομμύρια υπάρχει χρηματοδότηση blending από τότε που υπάρχει το σύστημα. Τι ποσοστό αντιπροσωπεύει αυτό. Δηλαδή τι ποσοστό χρηματοδοτείται από τα προγράμματα. 1,8 δις, τι σημαίνει αυτό. Και ποιο τμήμα σε σχέση με τα κονδύλια που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλη την αναπτυξιακή βοήθεια. Ποια είναι η σχέση αυτή. Δεν ξέρω αν ε, μπορώ να σας δώσω μια συγκεκριμένη απάντηση τώρα. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω είναι ότι το 1,8 δισεκατομμύρια αντιστοιχεί περίπου σε 800 εκατομμύρια βάση του Αναπτυξιακού Ταμείου και ένα δις είναι η χρηματοδότηση στα πλαίσια του προπολογισμού σε αυτό το 1 δισεκατομμύριο, 760 εκατομμύρια περίπου είναι για το Investment Facility και 250 εκατομμύρια χρηματοδοτήθηκαν στα πλαίσια του DCE στο Latin American Investment Facility, Asia Investment Facilities κλπ. 1,8 δις, λοιπόν, άδεμα πατάει η μνήμη μου, είναι ποσό που αντιστοιχεί σε 20 δις συνολικών επενδύσεων. 20 δις. Α, όχι, συγγνώμη, λάθος. 20 δισεκατομμύρια είναι επενδύσεις του δημοσίου τομέα από την Ευρώπη και αντιστοιχεί σε ένα συνολικό ποσό επενδύσεων 40 δισεκατομμυρίων. Ε, χοντρικά, εντάξει, σας δίνω χοντρικά γιατί πρέπει να τα επαληθεύσω πιο συγκεκριμένα. Τέλο αν δεν είναι 20 θα είναι 21 και αν δεν είναι 40 μπορεί να είναι 41, αλλά πάντως λίγο πολύ αυτή είναι η τάξη μεγέθους. Η χρηματοδότηση λοιπόν έγινε στα πλαίσια των προηγούμενων πολιτών δημοσιονομικών προοπτικών, αναπτυξιακή βοήθεια δηλαδή συν προπολογισμό συν φέντ. Το συνολικό ποσό ήταν περίπου 60 δισεκατομμύρια. 1,8 από την άλλη μεριά δισεκατομμύρια. Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε. Κατά τη γνώμη σας, τι είναι αυτό το οποίο οδηγεί στις επενδύσεις, που προκαλεί τις επενδύσεις, το γεγονός δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει στο blending βοηθάει ώστε οι άλλοι φορείς να δεσμευτούν και να χρηματοδοτήσουν είναι επειδή υπάρχει... Ελπίζω, ελπίζω λέει ο και της Επιτροπής. Ελπίζω και πιστεύω ότι επειδή εμείς δεσμευόμαστε και αναλαμβάνουμε κάποια υποχρέωση, ακολουθούν και οι υπόλοιποι οικονομικοί φορείς. Γι' αυτό εμείς πρέπει να βάλουμε δημόσιο χρήμα σε προγράμματα που χρηματοδοτεί ο δημόσιος τομέας αλλά και, η... και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν αποφασιστική σημασίας για δύο λόγους και αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε. Αποτελεί έναν οικονομικό μοχλό, δηλαδή το γεγονός ότι καταστήσαμε εφικτό να μειωθεί το κόστος γιατί τώρα μειώνεται το κόστος της επένδυσης, γιατί μειώνονται τα επιτόκια ή μειώνεται το συνολικό ποσό που πρέπει να δανειστεί η χώρα. Άρα μειώνεται το κόστος για τη δική χώρα. Είμαστε πεπισμένοι λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η μόχλευση και έτσι κάποιες επενδύσεις έγιναν δυνατές ακριβώς επειδή μειώθηκε το συνολικό κόστος της επένδυσης. Υπάρχουν τώρα άλλα προγράμματα για τα οποία θα ήθελα να φέρω εδώ κάποια διευκρίνηση. Ίσως να μπορούσε και πριν τη δικιά μας την επένδυση να γίνει ένα πρόγραμμα, αλλά επηρεάζουμε τον σχεδιασμό είτε όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ή τις κοινωνικές επιπτώσεις σε σχέση με ό,τι είχε προβλεφθεί στην αρχή. Άρα έτσι όπως αναλύουμε εμεί τα πράγματα, έτσι καλώς υπάρχει η ενδιάμεση αξιολόγηση, έτσι. Είτε για το Neighbor investment Facility, είτε για άλλα είναι σαφές ότι τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων αυτών μας λένε ότι υπάρχουν αυτού του είδους οι συνέπειες, επειδή μειώνεται το κόστος της επένδυσης είναι πιο εφικτές οι επενδύσεις, ή από την άλλη μεριά στην αρχή, στον σχεδιασμό προστίθενται κάποιες περιβαλλοντικές ή κοινωνικές προδιαγραφές. Αναρωτιέμαι για όλα αυτά. Πώς αξιολογείται το πρόγραμμα αυτό μέσα στην Κομισιόν, γιατί οι επενδύσεις που κάνουμε 1,7 δις σε ένα χρόνο, η Παγκόσμια Τράπεζα επενδύει ούτε και ξέρω σε πόσα φτάνει αλλά ε, φτάνει σε πολλαπλάσια, εκατοντάδες δις ετησίως. Και έχει ε, φανταστικά, φανταστικά ε, υπαλλήλους δίνει το 8% όταν δίνει το 8% εκτιμά πως έχει κάνει τα βασικά έχει κάνει δηλαδή την ε, περιβαλλοντική μελέτη, την μελέτη της σκοπιμότητας. Ποια είναι η προστιθέμενη αξία της Κομισιόν σε αυτό το τεράστιο μηχανισμό. Τα δικά μας προγράμματα εν γέννη, όπως και οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτεί Κομισιόν, καταρχήν παρουσιάζονται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που πρέπει να μας υποβάλουν τα προγράμματά τους ε, με ε, αναπαραίτητο τις ε, συνοδευτικές μελέτες που έχουν εκπονήσει ώστε να λάβουμε απόφαση. Στη συνέχεια τα προγράμματά μας προετοιμάζονται και αξιολογούνται δηλαδή σε ποιο βαθμό θα πρέπει να συμβάλλουμε αξιολογούνται όχι από την μικρή ομάδα που εγώ διαχειρίζομαι, αλλά από τους συνάδελφους των τεχνικών υπηρεσιών. Εξωτερικές υπηρεσίες, η εξωτερική υπηρεσία επίσης αξιολογεί και οι συνάδελφοι ε, που είναι στην αντιπροσωπεία. Ακολουθεί δηλαδή την πορεία που ακολουθεί οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα μέσα στην Κομισιόν. Το λόγο έχει η κυρία Γκέρες. Πρέπει να θέσω ακόμα μια ερώτηση. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ έχω μια ερώτηση κατανόησης. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά την τεχνική Ε, θα μου πείτε αν είναι η ανάλυση μου σωστή. Χρηματοδοτούμε ένα project με το μέσο αυτό blending σε μια αναπτυσσόμενη χώρα. Το πρόγραμμα αυτό κοστίζει 100 εκατομμύρια ευρώ. Τα 30 καταβάλλονται υπό μορφή ε, δωρεών και τα 70 εκατομμύρια κινητοποιούνται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Το ερώτημά μου είναι ποια δέσμευση η Κομισιόν ε, αναλαμβάνει απέναντι στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Είπατε ότι μειώνεται το κόστος του δανείου ή το κόστος του επένδυση. Μα τα δύο αυτά όμως δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εάν καταβάλλετε μια δωρεά της τέξου 30% καθιστάτε την επένδυση πιο προσιτή για τον επενδυτή. Στην περίπτωση του blending μπορείτε να καταβάλλετε χρήματα σε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που το επιτρέπει να πρημοδοτήσει το επιτόκια, τα επιτόκια. Συμβαίνει αυτό. Εάν κατάλαβα καλά, σας θέσω μια επιπλέον ερώτηση. Στην παρουσίαση που θα έχουμε τον Απρίλιο, μπορούμε επίσης να έχουμε τα επιτόκια που καταβάλλονται στο πλαίσιο της μικροχρηματοδότησης, γιατί εκεί δεν υπάρχουν πρημοδοτήσεις των επιτοκίων. Και είναι ένα ε, ε, ε, μέσο το οποίο χρησιμοποιείται για τους πιο φτωχούς. Ενώ ε, χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τις κεφαλαγορές, Τα προγράμματα αυτά όμως χρηματοδοτούνται από τις κεφαλαγορές τα υπόλοιπα και με επιτόκια πολύ ψηλότερα που φτάνουν το 11, 12 και μέχρι και 16% γιατί λοιπόν να γίνει αλλαγή των επιτοκίων για επενδύσεις που μπορεί να αποφέρουν εμπορικό όφελος ενώ αφήνουμε τους στοχότερους να, να χρηματοδοτηθούν με τις συνθήκες της αγοράς. Πράγμα το οποίο δεν καθιστά τη μικροχρηματοδότηση λιγότερο αποδοτική. Ίσως να οφείλεται αλλού ας πούμε, στην υπηρεσία τη συνοδευτική που πλησιώνει κάθε τέτοιο εγχείρημα, όπου υπάρχει παρακολούθηση των επενδύσεων που γίνεται διαρκώς. Πράγμα που καθιστά το κόστος των χρημάτων που καταβάλλεται στην μικρό χρηματοδότηση εξαιρετικά δαπανηρό, εξαιρετικά υψηλό είναι κάπως περίπλοκη η ερώτησή μου, αλλά πιστεύω πως με καταλάβατε. Με καταλάβατε? Ναι, βεβαίως. Μία απόχρωση ίσως ε, στο πώς μας παρουσιάσετε τα πράγματα. Το πρώτο είναι ότι συνήθως Δεν βάζουμε 30 εκατομμύρια για μια, χρηματοδότηση, μια επένδυση 100 εκατομμυρίων, βάζουμε πολύ λιγότερα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, έχετε απόλυτα δίκιο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις δύο, δύο τρόπους. Δηλαδή, μπορούμε να δώσουμε μια άμεση επιδότηση στο ο κράτος δικαιούχο, δηλαδή μειώνουμε το κόστος της επένδυσης γιατί χρειάζεται μικρότερη επένδυση ή μπορούμε να κάνουμε μια επιδότηση των επιτοκίων, άρα μειώνουμε το κόστος του δανείου διότι επιδοτούμε άμεσα τα επιτόκια. Και εδώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους δύο τρόπους. Μας επιτρέπεται από τον δημοσιονομικό κανονισμό, είτε δηλαδή δίνουμε άμεσα την επιδότηση στην τράπεζα και μειώνουμε έτσι τα επιτόκια, είτε το δίνουμε στον χώρα δικαιούχο και τα δύο αυτά προβλέπονται. Έχουμε μία ανεμπειρία και από τις δύο αυτές μορφές επιδότησης επιδότηση στα επιτόκια που γίνεται κυρίως στο πλαίσιο του African Investment Trust Fund, το οποίο το διαχειρίζεται η ΕΤΕΠΑ. Η Κομισιόν ε, συμβάλλει εκεί και εκεί έχουμε τη επιδότηση των επιτοκίων. Αυτό προτιμάει η ΕΤΕΠΑ Εμείς στις ε, διευκολύνσεις ε, για τις επενδύσεις ε, ε, χρησιμοποιούμε ε, τι άμεσε επενδύσει στι χώρε δικαιούχου, γιατί πιστεύουμε πως αυτό έχει πλεονεκτήματα στη διαχείριση από πλευράς τη Κομισιόν γιατί άμεσα μειώνεται το κόστος τη επένδυση. Αλλά έχετε δίκιο ότι προβλέπονται και τα δύο αυτά. Προσπαθούμε να έχουμε ένα εφέ μόχλευσης μεγαλύτερο ενώ εσείς μιλήσατε για το 1 τρίτο. Ενώ εμείς έχουμε μόχλευση ανάμεσα στα 10 και 20. Κύριε Γκέρενς, πρέπει να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί είναι πολύ συναρπαστική, αλλά έχουμε και άλλα να μελετήσουμε. Νομίζω πως τα μέλη της Επιτροπής δεν καταχρώνται του χρόνου ομιλία του σήμερα. Euh, l'instrument de financement. Εάν έχετε λοιπόν χρησιμοποιήσει το μέσο χρηματοδότησης, εάν παρέμβετε στο κόστος των χρημάτων και αν αυτό αποτελέσει συνήθεια, μήπως δεν θα ήταν φαύλο το αποτέλεσμα, δηλαδή τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αυξάνουν τα επιτοκιά τους διότι ούτως ή άλλως ξέρουν ότι θα μειωθεί το επιτόκιο χάρη στην συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του blending. Δηλαδή το σύστημα είναι αρκετά ασφαλές ώστε να προληφθεί αυτό. Ναι βεβαίως, βεβαίως. Είναι ένας κίνδυνος και είναι κάτι για το οποίο πρέπει να επαγρυπνούμε για αυτή τη συζήτηση του blending υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι όπως αυτός που αναφέρατε. Υπάρχει και ένας δεύτερος κίνδυνος που μπορώ αμέσως να σας τον πω. Δηλαδή οι χώρες εταίροι να ε, χρεωθούν υπερβολικά διότι μπορούν να πάρουν χρήματα σε τιμές χαμηλότερες από ό,τι αν δεν επιδοτούνταν. Είναι δύο πτυχές λοιπόν όπου πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ ώστε να εξασφαλίζουμε ότι ενώ θα μπορέσει να υλοποιηθεί η επένδυση και θα εξασφαλιστούν οι πόροι, να μην προκαλούμε στρεβλώσεις της αγοράς ή τεχνητή αύξηση των επιτοκίων για τις χώρες εταίρους. Αυτό φυσικά εξαρτάται και από την λειτουργία της αγοράς της ίδιας, γιατί οι χώρες δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα, κυρίως οι χώρες που μπορούν να ανατρέξουν σε διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης, θα έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν τις διάφορες προσφορές και να επιλέξουν εκείνη που έχει τα περισσότερα πλανεκτήματα. Η αλλαπάντησή μου είναι ναι, είναι ένα κίνδυνο και ένα κίνδυνο τον οποίο έχουμε υπόψη μας και παρακολουθούμε κάθε φορά προσεκτικά σε κάθε επένδυση. Πρόεδρος η Επιτροπή Ανάπτυξης θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί με προσοχή αυτό το μέσο. Αυτά. Ε, παρνάμε τώρα στο σημείο 11 της ημερήσιας διάταξης, όπου έχουμε την τρίτη και τελευταία μελέτη που παρουσιάζεται ενώπιον της Επιτροπής μας. Πρόκειται για μια μελέτη που αφορά τον αντίκτυπο των εμβασμάτων των μεταναστών στην οικονομία των αναπτυσσόμενων χωρών, των χωρών προέλευσής τους δηλαδή. Είναι αμέσως το λόγο στους συντάκτες της μελέτης, ώστε να μας παρουσιάσουν τα βασικά της στοιχεία. Κυρία, κυρία Κάριν Λουμπάντου, έχετε το λόγο. Merci bien pour euh, la parole. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας παρουσιάσω στα αγγλικά την μελέτη, μια που έγινε στα αγγλικά η μελέτη και μετά στα γαλλικά θα συνεχίσω για να απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιάσω τα βασικά ευρήματα της ε, έκθεσης για τον αντίκτυπο των εμβασμάτων στις ανατσόμενες χώρες. Βεβαίως ε, μελετάμε το τι γίνεται σε μικρό και μακρό επίπεδο, το θέμα της αγοράς εμβασμάτων, τα βασικά ζητήματα χρήσης των εμβασμάτων για σκοπούς ανάπτυξης, το τι γίνεται με την ατζέντα για μετά το 2015 και τον πιθανό ρόλο που θα μπορούσαν να παίξουν τα εμβάσματα στην ατζέντα μετά το 2015 και τέλος οι συστάσεις μας. Όπως είπα, ο στόχος ήταν να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο των εμβασμάτων. Κάποιοι περιορισμοί αφορούν την έλλειψη δεδομένων στις αναπτυσσόμενες ε, χώρες. Αν δει κανείς ε, τη βιβλιογραφία που υπάρχει, ε, ήταν κάποια έρευνα γραφείου της ήδη φυστάμενης έρευνας και όχι άμεση αξιολόγηση επιτόπου ε, και βέβαια υπήρχαν ε, και περιορισμοί χρονικοί. Οπότε τα βασικά ευρήματα σε μικρό και μακρό επίπεδο ε, είναι πως υπάρχουν και θετικές και αρνητικές πτυχές αναψώμενες χωρίς στο μικρό επίπεδο δηλαδή στο επίπεδο του νοικοκυριού, του ατόμου, ο θετικός αντίκτυπος είναι να βοηθηθούν οι οικογένειες να ικανοποιήσουν τις βασικές τους ανάγκες και να έχουν έτσι περισσότερο εισόδημα για επενδυτικούς σκοπούς. Από την άλλη, αρνητική πτυχή είναι το εξής, ότι αυξάνονται οι τιμές οι τοπικές ε, της γης, ε, κατασκευαστικών υλικών ε, και άλλων αγαθών στην τοπική οικονομία. Ένα άλλο αρνητικό των εμβασμάτων αφορά τις ανισότητες μεταξύ νοικοκυριών που λαμβάνουν και δεν λαμβάνουν εμβάσματα. Και βεβαίω ε, ένα άλλο ζήτημα είναι πως ε, υπάρχει μία εξάρτηση και βεβαίως ασκείται και μία πίεση προς αυτούς που στέλνουν τα λεφτά. Έτσι. Δηλαδή πολλοί σκέφτονται πως αυτοί που στέλνουν τα λεφτά είναι μετανάστες, αλλά δεν συμβαίνει πάντα αυτό. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε άλλος. Είναι δηλαδή μια πίεση ε, μετανάστε στη χώρα προορισμού. Στο μικροεπίπεδο έχουμε θετικό αντίκτυπο κυρίως όσον αφορά το εθνικό εισόδημα, εάν μεταφέρονται από επίσημους διάβλους και μια άλλη θετική πτυχή είναι πως ε, προωθείται έτσι η τοπική οικονομία με το να προωθείται η επένδυση στο τοπικό επίπεδο. Τα αρνητικά στο μακροεπίπεδο είναι πως υπάρχει ανατίμηση του νομίσματος με αρνητικές συνέπειες για τις εξαγωγές, αύξηση του πληθωρισμού και κάποιες ανισότητες ε, μεταξύ των περιοχών που λαμβάνουν και αυτών που δεν λαμβάνουν εμβάσματα. Βασική πτυχή επίσης είναι το ότι τα εμβάσματα μπορούν να συνεισφέρουν στην ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών που κανονικά θα έπρεπε να είναι δημόσιες. Οπότε η πτυχή αυτή οπωσδήποτε βασίζεται στις υφιστάμενες υποδομές στο τοπικό επίπεδο. Παραπέρα. Τώρα θα ήθελα να αναφέρω πως ε, εργάζομαι στο ζήτημα της ε, στο τμήμα του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στην ε, Γενέβη που αφορά τις εργασιακές σχέσεις. Λοιπόν, η αγορά αυτή των εμβασμάτων υπάρχουν επίσημοι και άτυποι διάβλοι οι επίσημοι δίωδοι αφορούν την ασφάλεια, την αξιοπιστία, υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές και βεβαίως να εμβαθυνθεί η ο βαθμός δημοσιονομικής ε, διαμεσολάβησης της χώρας. Και βέβαια υπάρχει το ζήτημα των ειδότησης και οι νέες ε, τεχνολογίες ε, που βοηθούν. Βεβαίω, το πρόβλημα εδώ πέρα είναι πως δεν υπάρχει διαφάνεια και ανταγωνισμός, υπάρχουν αποκλειστικές συμφωνίες Ε, μεταξύ τραπεζών και τέτοιων εταιριών και οι αποκλειστικές αυτές συμφωνίες περιορίζουν ε, τον ε, ανταγωνισμό. Επίσης υπάρχουν περιορισμένες υποδομές στις αναπτυσσόμενες χώρες, υπάρχει το περίπλοκο ρυθμιστικό περιβάλλον, αυτό αφορά συγκεκριμένα της, ε, την ε, οδηγία καταπολέμησης ε, του εγκλήματος και της τρομοκρατίας που βεβαίως δημιουργεί κάποιες προκλήσεις για τις αναπτυσσόμενες χώρες και παραδείγματος χάρη το είδαμε αυτό πρόσφατα με το κλείσιμο των επισήμων διάβλων στην Σομαλία με την Barclays η οποία έκλεισε κάποιες τέτοιες εταιρείε. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα για τις, ε, τους επίσημους διαβούλους αφορά τη μη πρόσβασιμότητα για τους μετανάστες χωρίς έγγραφα που δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες τέτοιες ε, στις χώρες ε, προορισμού και όσον αφορά όπως είπαμε τα άτυπα μέσα αυτά θεωρούν κάποιοι πως θα μπορούσαν να αποτελέσουν ε, πιθανό μέσο τρομοκρατικών, ε, τρομοκρατικής χρηματοδότησης. Δεν συμβαίνει αυτό πάντα. Τα άτυπα μέσα θα μπορούσαν να έχουν παραδείγματος χάρη αιτία την κρίση στις περιοχές αυτές. Οπότε, εδώ πέρα έτσι γρήγορα, μπορούμε να έχουμε μια κάποια προσέγγιση ε, που θα κάνει κάποιες διακρίσεις όσον αφορά την χρηματοδότηση τρομοκρατίας, εγκλήματος κτλ. Όπως είπα, τα βασικά ζητήματα είναι η διαφάνεια, η έλλειψη τοπικής υποδομής, ε, η έλλειψη ανταγωνισμού, κυρίως στους διάβλους από νότο προς νότο, όπου το κόστος μπορεί να είναι και πάνω από 15% του ποσού που εμβάζεται. Το δύσκολο ρυθμιστικό περιβάλλον, όπως και η έλλειψη συλλογής ε, δεδομένων για το τι μπορεί να γίνει σε αυτές χώρες. Οπότε, έχουμε εδώ πέρα το τι γίνεται με το τι μπορεί να γίνει με τη μόχλευση των εμβασμάτων. Αυτά έχουν επιλεγεί τα έργα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο κράτους μέλους και στο διεθνές επίπεδο. Έχουν συγκεντρωθεί από διαφορετικέ κατηγορίες, από την εναρμόνιση συλλογής δεδομένων ε, για τα εμβάσματα και βεβαίως ε, από την εναρμόνιση των μεθόδων αυτών βελτίωση των διάβλων νότου-νότου. Επίσης έχουμε εδώ πέρα συγκεντρώσει όλα τα έργα που έχουν εφαρμοστεί. για να εκμεταλλευτούν περισσότερο δυνατό, τις δυνατότητες που δίνουν τα εμβάσματα. Επίσης η βελτίωση της σχετικής αγοράς, π.χ. η τραπεζική μέσω κινητών είναι ένας πάρα πολύ καλός τρόπος για να μειωθεί το κόστος των εμβασμάτων. Τα εμβάσματα επίσης και τα σχετικά προϊόντα όπως παραδείγματο χάρη η οικονομική έτσι, στοιχειώδης οικονομική εκπαίδευση και άλλα ζητήματα που αφορούν π.χ. τη χρηματοδότηση του κλίματος και βεβαίως ε, δύο βασικοί τομείς ε, εδώ πέρα μας ανησυχούν, κυρίως ε, η πρόσβαση μεταναστών χωρίς έγγραφα σε επίσημους διάβλους και το τι κάνει αυτός ο κανονισμός για τις τιμές στις χώρες της ε, έχουμε λοιπόν μία διαφάνεια για την ατζέντα μετά το 2015 και τον πιθανό ρόλο των εμβασμάτων. Η σχέση μεταξύ εμβασμάτων και άλλων πηγών εισοδήματος ε, στις αμψόμενες χώρες. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, αυτά είναι τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, ή τα εμβάσματα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πηγή εξωτερικής χρηματοδότησης σε αυσόμενε χώρες μετά την αναπτυξιακή βοήθεια και τις άμεσες ξένες επενδύσεις και πολλές μελέτες έδειξαν πως τα εμβάσματα άντεξαν κατά τη διάρκεια της κρίσης, πάντα σύγκριση με τις άλλες ροές. Οπότε επίσης υπάρχει η δυνατότητα να προσφέρουν κάτι στην ανάπτυξη, αλλά ταυτόχρονα είναι ε, ιδιωτικά χρήματα των μεταναστών. Και όλες οι πολιτικές που θέλουν ε, να εκμεταλλευτούν αυτά τα εμβάσματα πρέπει πρώτα απ' όλα να σκέφτονται τα δικαιώματά τους και τις ανάγκες τους. Έτσι, γιατί είναι τα δικά τους ιδιωτικά χρήματα. Και ένα άλλο θέμα βέβαιος είναι πως δεν μπορεί να θεωρηθούν ως υποκατάστατο της ε, ξένης αναπτυξιακής βοήθειας ή των άμεσων ξένων επενδύσεων. Επίσης, οι εθνικοί λογαριασμοί, τα εθνικά εισοδήματα έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν στην ανάπτυξη των χωρών αυτών. Τώρα για να πάμε κάπως πέρα από το ζήτημα της παρακολούθησης, ένα άλλο ζήτημα είναι και η ευημερία των μεταναστών υπό την έννοια πως βλέπουμε εδώ πέρα πως ε, πάρα πολλοί κόσμος θέλει να εκμεταλλευτεί αυτά τα εμβάσματα, αλλά πρέπει να σκεφτούμε και την ποιότητα ζωής τους στις χώρες προορισμού, πώς θα μπορέσουν να βοηθήσουν τις χώρες προέλευσής τους ε, και στην ανάπτυξή τους, εάν στη χώρα προορισμού δεν έχουν ε, καλές συνθήκες ζωής. Τελευταία διαφάνεια αφορά συστάσεις και ιδέες. Από ό,τι κατάλαβα... Είδαμε τον ε, διεθνή διάλογο. Το πρώτο το οποίο πρέπει να γίνει είναι να δούμε τα εμπόδια που υψώνονται από τους κανονισμούς μεταφοράς ε, χρημάτων. Αυτό αφορά πάρα πολύ την αγορά των εμβασμάτων και οι μικρές ε, τέτοιες εταιρείες κλείνουν. Οπότε αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα, βασικές συστάσεις ε, για τα ζητήματα αυτά που απορρέουν από τον σχετικό κανονισμό. Το δεύτερο είναι πως πρέπει να εναρμονιστούν ε, τα εμβάσματα, οι συλλογές δεδομένων και καθορισμού των εμβασμάτων, γιατί διαφορετικές χώρες λέγουν διαφορετικά δεδομένα και είναι δύσκολο να γίνει κάποια σύγκριση, γιατί ακριβώς η διαδικασία συλλογής ε, δεν είναι ακριβώς ίδια. Ε, μια άλλη βασική σύσταση αφορά την συνεργασία με την διασπορά και να υπάρξει μια καλύτερη αντίληψη και ενσωμάτωση των μεταναστών στην χώρα υποδοχής και βεβαίως να αντιληφθούμε το γιατί, το ποια είναι τα εμπόδια όσον αφορά το γιατί δεν θέλουν να επενδύσουν οι μετανάστες στην ε, χώρα προέλευσης τους. Ε, ένα άλλο βασικό ζήτημα είναι να επιτευχθεί η συνεργασία στον τομέα του Νότου και να υπάρξει μια συνοχή στην πολιτική, για να υπάρξει καλύτερη, νομίζω, καλύτερος αντίκτυπος και συνεργασία μεταξύ των διαφόρων αυτών τομέων και άλλη μια σύσταση είναι να σχεδιαστούν κατάλληλα κίνητρα και πολιτικές. Αυτό αφορά τη μείωση του κόστου συναλλαγής, ένα βασικό ζήτημα που θα μπορούσαν να κάνουν οι πολυμερείς φορείς και βεβαίως να μην φορολογούνται τα εμπάσματα, όπως ξέρουμε πως κάνουν κάποιες χώρες στις χώρες προέλευσης αλλά και στις χώρες ε, προορισμού. Ε, πρέπει να αποφευχθεί αυτό για να υπάρξει μεγαλύτερο αναπτυξιακό δυναμικό. υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, δηλαδή δεν είναι ξένα κονδύλια ούτε διεθνής βοήθεια τα εμβάσματα, αλλά θα μπορούσαν μετά το 2015 να θεωρηθούν κάτι τέτοια, όπως είπα, σεβόμενοι πάντα τα δικαιώματα των μεταναστών. Και τέλος, η βελτίωση των εθνικών υποδομών σε αναπτυσσόμενες ε, χώρες. Η ανάπτυξη είναι ευθύνη των εθνικών αρχών και όχι των μεταναστών. Αυτό είναι βασικό. Ακόμα και οι πολιτικές στοχεύουν τα εμβάσματα είναι καλές εάν οι υποδομές στο εθνικό επίπεδο όμως δεν αναπτυχθούν, δεν υπάρχει κάποιο όφελος. Έτσι δηλαδή δεν θα ωφεληθεί ο τοπικός πληθυσμός. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Oui, euh, Ευχαριστώ πολύ για αυτές τις τόσο ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι το υπερβολικό κόστος στις μεταφορές αυτές χρημάτων, στα εμβάσματα, το κόστος δηλαδή που καλούνται να πληρώσουν οι οικογένειες ε, αυτές που βρίσκονται στη χώρα προέλευσης. Τι είναι αυτό που εξηγεί το υπερβολικό αυτό κόστος. Είναι το θέμα της συναλλαγής, της... Ε, πρέπει να δούμε τη διαφορά του κόστους ανάμεσα ε, στα ποσά που μεταφέρονται ε, βάσει του φράγκου που έχει να κάνει με το ευρώ, που συνδέεται με το ευρώ παρά από τις χώρες εκείνες, το ΣΕΦΕΑ. Μπορείτε λοιπόν να μας δώσετε παραπάνω εξηγήσεις, να μας δώσετε μια εικόνα για να καταλάβουμε τι γίνεται με την σταθερότητα από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δυτικής Αφρικής. Και δεύτερη ερώτηση, όταν τα χρήματα μεταφέρονται από μια χώρα του Βορρά σε μια αναπτυσσόμενη χώρα. Σε ένα λογαριασμό, σε μια τράπεζα που είναι θυγατρική τράπεζα για παράδειγμα. Το κόστος είναι το ίδιο τότε ή είναι χαμηλότερο. Η Μπεν Πεμπαριμπά για παράδειγμα, στην Μπουργκίνα Φάσο, ζητάει το ίδιο κόστος για την μεταφορά αυτή. Το ίδιο με τη μεταφορά σε μια άλλη αφρικανική ας πούμε τράπεζα. Έχω την εντύπωση δηλαδή ότι εδώ υπάρχει ένας παρασιτισμός γύρω από τις δραστηριότητε αυτές, από την οποία ζημιώνονται και αυτοί που στέλνουν τα χρήματα και αυτοί που τα λαμβάνουν. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα. Η κυρία Βάιντοβαν, παρακαλώ. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς για τη μελέτη, γιατί πιστεύουμε ότι έρχεται την κατάλληλη στιγμή μετά από την επέκταση του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση. Σημεριζόμαστε τα συμπεράσματα της μελέτης αυτής. Υπάρχει πρόοδος, αλλά μένουν πολλά να γίνουν στον τομέα των εμβασμάτων. Το συμπέρασμα αυτό υπογραμμίστηκε και στη μελέτη του 2012 που εκπώνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρουσιάστηκε και εδώ. Χαιρόμαστε πολύ επίσης για τη σημασία που δίνει η μελέτη στο θέμα των εμβασμάτων, ότι δεν πρέπει να θεωρηθεί ένα επιπλέον μέσος, μέσον μάλλον για ανάπτυξη, αλλά ότι είναι ένα συμπλήρωμα και χαιρόμαστε επίσης που η μελέτη δεν περιορίζεται στα θετικά των εμβασμάτων, αλλά αναγνωρίζει και τις δυνητικά αρνητικές επιπτώσεις. Συμφωνούμε με τις συστάσεις επίσης της μελέτης αυτής, γιατί ευθυγραμμίζονται με τη δικιά μας την προσέγγιση και συμφωνεί με τη δουλειά που κάνουμε εμεί όσον αφορά τα εμβάσματα σε αναπτυσσόμενε χώρες. Όπως γνωρίζετε, ίσως από το 2005 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει συγκεκριμένες δεσμεύσει στον τομέα των εμβασμάτων. Υπογραμμίζουμε την ιδιωτική φύση των εμβασμάτων και στόχος παραμείνει να προωθήσουμε πιο φτηνά εμβάσματα τα οποία να φτάνουν πιο γρήγορα στον προορισμό τους. Υπάρχουν κάποιες αλλαγές, υπάρχει κάποιος κατακαιρματισμός μερικές φορές που πλήττει τη συνοχή της πολιτικής, όπως η κυρία Λουμπάμπου ήδη είπε. Για παράδειγμα, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα εμβάσματα αποτελούν μέρος της ατζέντα για την μετανάστευση και την ανάπτυξη, αλλά αποτελούν μέρος και του ρυθμιστικού πλαισίου της εσωτερικής αγοράς και συνδέονται επίσης και με τις ρυθμίσεις κατά της τρομοκρατίας ή κατά της νομοποίησης παράνομου χρήματος. Όλα αυτά βέβαια έχουν κάποιες επιπτώσεις και αρνητικές μερικές φορές. Πρώτα απ' όλα δεν ε, πιστεύουμε πλήρως στην ατζέντα για τα εμβάσματα και υπάρχουν και θέματα συνοχής πολιτικής. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιλαμβανόμαστε τις προκλήσεις αυτές και προσπαθούμε να ενισχύσουμε τον συντονισμό μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συγχρηματοδοτήσει κάποιες από τις εμβληματικέ πρωτοβουλίες στον τομέα των εμβασμάτων, όπως την οικονομική διευκόλυνση για τα εμβάσματα και το Αφρικανικό Ινστιτούτο για τα εμβάσματα. Αξίζει εδώ επίσης να αναφέρουμε ότι η Financial Facility για τα ξεκίνησε με ευρωπαϊκή συνεισφορά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έφτασε στα 28 εκατομμύρια δολάρια με 100 εκατομμύρια συγχρηματοδότηση από άλλες οργανώσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης θα συνεχίσει να στηρίζει πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο να ενισχύσουν τον ανταγωνισμό στην αγορά την αφρικανική εμβασμάτων. Θα επιτρέψει στα αφρικανικά ταχυδρομεία, για παράδειγμα, να προσφέρουν περισσότερες οικονομικές υπηρεσίες στις οικογένειες των μεταναστών. Όσον αφορά τώρα τις μελλοντικέ μας προτεραιότητες, πιστεύουμε ότι πρέπει να δώσουμε περισσότερη προσοχή σε δύο τομείς που αναφέρονται μάλιστα στην τρέχουσα μελέτη. Πρώτον, κοινωνικές επιπτώσεις και δεύτερον, νομοθεσία. Η συζήτηση μέχρι τώρα έχει επικεντρωθεί πάρα πολύ στις θετικές πτυχές των εμβασμάτων. Στέκεται στις επιπτώσεις. Οι επιπτώσεις Τόσες όμως στις οικογένειες και στις κοινότητες της χώρες προέλευσης μπορεί να είναι τόσο θετική όσο και αρνητική. Τα εμβάσματα δεν αντικαθιστούν άλλα μέσα κοινωνικής προστασίας, ούτε αφαιρούν την ευθύνη από τις χώρες μέλη για να προσφέρουν τις κατάλληλες υπηρεσίες και πολιτικές. Για να μειωθούν οι αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις των ευασμάτων πρέπει να ενισχυθεί η συνειδητοποίηση όλων των πλευρών στις δυνητικά αρνητικές επιπτώσεις, έτσι ώστε να υπάρχει κατάλληλη νομοθεσία και να γίνονται παραγωγικές επενδύσεις. Η δεύτερη διάσταση στην οποία σκοπεύουμε να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στο μέλλον, έχει να κάνει με τα εμβάσματα νότου-νότου. Ανάμεσα στα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τα μέσα εξωτερικής συνεργασίας δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στα εμβάσματα αυτά νότου-νότου. Πολλά ακόμα μένουν να γίνουν για να βελτιωθεί η διαφάνεια πρώτα απ' όλα και ο ανταγωνισμός για τέτοιες μεταφορές εμβασμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για να αναπτύξει ακόμα περισσότερο την πτυχή αυτή στο μέλλον και ιδιαίτερα όπως υπογραμμίζει και η μελέτη στα πλαίσια της εποχής μετά το 2015. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε. Για τρία λεπτά τώρα το πολύ ο κύριος Φλωριάν Κράκ που μας κάνει την τιμή να είναι πάντα εδώ από το CDPM. Σας ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πολύ και πάλι που μου δίνετε το λόγο και ευχαριστώ και την κυρία Λουμπάμπο για την ε, τόσο πλήρη μελέτη που μας παρουσίασε όσον αφορά τις επιπτώσεις των ευασμάτων. Έχω τέσσερα σημεία μετά τις εξαίρετες συστάσεις και να προσθέσω και κάποιες. Πρώτον, όπως είπαν και άλλοι ομιλητές, είναι ιδιωτικό μέσο τα εμβάσματα. Συνεπώς, δεν έχουν σαν στόχο να στηρίξουν τους εθνικούς αναπτυξιακούς στόχους. Είναι ιδιωτική η φύση τους και δεν πρέπει κατευθείαν να πηγαίνουν στους αναπτυξιακούς στόχους. Οι συνάδελφοί μου και εγώ πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό οι ίδιες πολιτικές που στηρίζουν την αναπτυξιακή πτυχή των ε, εμβασμάτων δημιουργούν και πεδίο για επενδύσεις. Πρέπει να υπάρξει εμπιστοσύνη, να δημιουργείται δηλαδή ένα κλίμα εμπιστοσύνης για επιδέσεις, να υπάρχει κοινωνική σταθερότητα και να μην αγνοούμε τα εμπόδια που υπάρχουν στις επενδύσεις πολλές φορές στις αναπτυσσόμενες χώρες. Έπειτα, τα νοικοκυριά δεν αποφελούνται με τον ίδιο τρόπο από τα εμβάσματα. Πρώτα απ' όλα, γιατί δεν έχουν όλα τα νοικοκυριά κάποιο μετανάστη να στέλνει εμβάσματα. Υπάρχουν πιο πλούσια νοικοκυριά και άλλα λιγότερο. Οπότε ίσως θα πρέπει να δούμε και το κόστος της μετανάστευσης και πώς θα μειωθεί αυτό και στην ατζέντα για μετά το 2015 να ένας τομέας που θα έπρεπε να προσεχτεί περισσότερο, να μην ασχοληθούμε μόνο με το κόστος των εμβασμάτων, αλλά το γενικότερο κόστος της μετανάστευσης. Έπειτα να δούμε τη σχέση των εμβασμάτων με την ανάπτυξη. Ακούστηκε η σχέση αυτή πολλές φορές εδώ. Και εμείς το έχουμε διαπιστώσει και πρέπει να υπάρξει μια καλή ισορροπία ανάμεσα στις διάφορες πολιτικές. Είπαμε ότι έχουμε ε, την καταπολέμηση της νομιμοποίησης παράνομου χρήματος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν έχει αναλάβει δεσμεύσεις όπως και η G8 και η G20, αλλά λίγα έχουν γίνει μέχρι τώρα. Παράδειγμα, ο στόχος για τη μείωση του κόστους των εμβασμάτων 5% μέχρι το 2014. Είμαστε στο 2014 και νομίζω ότι το κόστος των εμβασμάτων είναι κάπου 10% και υπάρχουν και ψηλότερα. Η μελέτη πάντως δείχνει ότι πολλές χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κάνει κάποια πρόοδο. Οπότε γιατί έχουμε αποτύχει μέχρι τώρα. Τέλος, κάπως πιο αφηρημένα. Κάτι που δεν είδα να αντικατοπτρίζεται στην έκθεση αυτή στη μελέτη είναι ότι η τυποποίηση ίσως να μην είναι και καλύτερη λύση για τα εμβάσματα. Όλες οι συστάσεις μιλάνε για τυποποίηση της μεταφοράς εμβασμάτων. Όμως πρέπει έτσι κι αλλιώς να διατηρήσουμε και τα θετικά των άτυπων εμβασμάτων. Κάποιος ρώτησε πώς ξέρουμε ότι οι τράπεζες ή οι άλλες οι εταιρείες που κάνουν αυτή τη μεταφορά εμβασμάτων κατά πόσο είναι κατάλληλες, πώς μπορεί κανείς να το ξέρει. Πρόεδρος, έχουμε καθυστερήσει, λυπάμαι. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Λουμπάμπου για να ολοκληρώσει. Σύντομα παρακαλώ, το πολύ τρία λεπτά έχετε στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα. Πολύ σύντομα για να απαντήσω στο ερώτημα, στο θέμα του κόστους. Είναι αλήθεια, όπως είπα, ότι υπάρχουν καταχρηστικές συμφωνίες ανάμεσα σε εταιρείε με μεταφοράς χρημάτων και τις ε, τοπικές τράπεζες που στην ουσία έχουν πάρει το 70 με 75% της αγοράς. Είναι αλήθεια το να χρησιμοποιήσει κανείς τους επίσημους ε, ε, διόδους είναι πραγματικά αρνητικό. Και αν μπορώ να σας πω για τη δική μου εμπειρία, είναι σαφές ότι η ιδέα της τυποποίησης και πάλι για να μιλήσουμε αυτό, για αυτό που σήμερα λέμε financial inclusion, δηλαδή να καταστούν οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες προσιτές στους ανθρώπους των αναπτυσσόμενων χωρών, αλλά ταυτόχρονα οι μεταφορές, τα εμβάσματα που γίνονται άτυπα, εγώ και εγώ χρησιμοποιώ αυτές τα εμβάσματα τα άτυπα, διότι το να μπορεί κανείς να στείλει χρήματα και να δει το 15% των χρημάτων που στέλνουμε να πηγαίνει στις ε, εταιρείε των εμβασμάτων είναι ε, τεράστιο ποσοστό. Οπότε δεν μπορούμε να συμβάλλουμε με αυτόν τον τρόπο στην ανάπτυξη των χωρών ε, προέλευσης. Ένα άλλο σημείο το οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως από το πρώτο, η πρώτη ερώτηση ήταν νομίζω, αν μπορούμε να δώσουμε ένα γράφημα με περισσότερες λεπτομέρειες ε, όσον αφορά το κόστος. Ναι, αυτό μπορούμε να το κάνουμε, οπότε μην διστάσετε να... Ίσως και μέσως μετά από αυτή την συνεδρίαση να μου το ξαναθυμίσετε για να σας το στείλω. Για τις τράπεζες, από εκεί ξεκινάει και η ιδέα εντοπισμού νέων ε, δρόμων ε, για μεταφορά χρημάτων, ας πούμε η ε, κινητή τραπεζική, όπως στην περίπτωση της Κένιας, αλλά και πάλι η βασική ευθύνη επιβαραίνει την ε, τοπικές αρχές γιατί το MPSA που είναι η χρήση της κινητής τηλεφωνίας αν ε, πήρε τόσο μεγάλες διαστάσεις είναι επειδή οι εθνικές αρχές ήταν υπέρ αυτού του σχεδίου και μέσω της κινητής τηλεφωνίας μειώθηκε το κόστος ε, των εμβασμάτων. Πρέπει να δούμε δηλαδή ποιες υποδομές υπάρχουν σε κάθε χώρα ώστε να δούμε ποιο είναι το δυναμικό των ε, εμβασμάτων και πώς αυτό μπορεί να μεγιστοποιηθεί χάρη στις ε, καινούργιες τεχνολογίες. Γι' αυτό και είναι τόσο σημαντικές καινούργιες τεχνολογίες για την Αφρική. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ τέλος για αυτή τη μελέτη που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και που θα μας εμπνεύσει και στην επόμενη θητεία. Τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης σήμερα και μας μένουν 35 λεπτά για να το συζητήσουμε. Και αυτό έχει σχέση με τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την παγκόσμια σύμπραξη για αποτελεσματική αναπτυξιακή συνεργασία. Κατά τη διάρκεια του φόρμα ανωτά του επίπεδου για την αποτελεσματικότητα της ενίσχυσης που θα γίνει στο Μεξικό τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους. Όπως γνωρίζετε, το πρόγραμμα για την αποτελεσματικότητα της ε, ε, αναπτυξιακής συνεργασίας ε, προκύπτει από την συνένεση του Μοντερή του 2002. Πρόκειται για μια σειρά από φόρα που έχουν συνεδριάσει στην Ρώμη το 2003, στο Παρίσι το 2005, στην Άκρα το 2008 και τέλος το 2011. Ε, θέλουμε να φτιάξουμε ένα νέο είδος εταιρική σύμπραξης για την ανάπτυξη όπου θα συμμετέχουν όλα τα συμβαλόμενα μέρη του αναπτυσσόμενου κόσμου. Ε, δεν αρκεστήκαμε στο να επιβεβαιώσουμε τις προηγούμενες δεσμεύσεις αλλά δεσμευτήκαμε για την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας η πρώτη συνεδρίαση της ε, Παγκόσμιας Σύμπραξης για την Αποτελεσματικότητα της ε, ε, Απτυξιακή Βοήθειας στο Μεξικό είναι ένας τρόπος για να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα του προγράμματος καθώς και τη διάρκεια του μετά το 2015. Και δίνω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον κύριο Μαρτέν Πράντα, για 7 λεπτά. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όντως, η υπουργική διάσκεψη του Μεξικό είναι πολύ σημαντική για το μέλλον της ε, σύμπραξης που δημιουργήθηκε στο Βουσάν. Και αυτό γιατί πιστεύουμε πως η αξιοπιστία όλου του χειρήματος ε, διακυβεύεται σας ε, πω σύντομα τι περιλαμβάνουν τα πορίσματα του Συμβουλίου για να δούμε τι μπορέσαμε να φτιάξουμε μετά το Τουσάν και ποια είναι τα αποτελέσματα δηλαδή για την ώρα. Θα έλεγα λοιπόν ότι από την πλευρά των θετικών αποτελεσμάτων πρέπει να υπογραμμίσουμε την ένταξη του παγκοσμίας σύμπραξης του ΤΟΣΑΝ, μια αποτελεσματικότητα και συμπερίληψη ένταξη που δεν ε, περιορίζεται στους παραδοσιακούς δωρητές αλλά και ε, συμπεριλαμβάνει και τους νέους δωρητές αναδυόμενες χώρες αλλά και επίσης εκπροσώπους εκπροσώπους τη κοινωνίας των πολιτών, του ιδιωτικού τομέα, διαφόρων κοινοβουλίων, τοπικών αρχών και ιδρυμάτων. Πρόκειται για μια πλατφόρμα πραγματικά ευρεία και αυτό είναι θετικό και για τις μελλοντικές συζητήσεις για το πλαίσιο ανάπτυξης μετά από το 2015. Υπάρχει άλλο ένα θετικό στοιχείο και αυτό αντικατοπτρίζεται και στην ατζέντα της Υπουργικής ότι υπάρχουν νέα θέματα όπως η κινητοποίηση των ε, χώρων εσόδων, ο ρόλος των ιδιωτών αλλά και η συνεργασία βορανότο που αποκτούν όλα ένα και μεγαλύτερη προτεραιότητα στην αναπτυξιακή κοινότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πολύ Αυτηρή όμως σε αυτό ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε τις δεσμεύσει που προέρχονται από αυτέ τι διάφορε διασκέψει, Παρίσι, Άκρα, όσον αφορά την αποδοτικότητα της ενίσχυση, γιατί Ακόμα κι αν η αναπτυξιακή βοήθεια σε σύγκριση με εσωτερικού πόρους είναι περιορισμένη, έχουμε δεσμεύσει και είναι σημαντικό να δείξουμε ότι τι εφαρμόζουμε. να δείξουμε ότι μπορεί να έχουμε δηλαδή αποτελέσματα και μετά από το, τούσαν ΣΑΝ. Ε, σημαντική είναι η δέσμευση των αναπτυσσόμενων χωρών, Κίνα, ε, Ινδία, Βραζιλία έτσι ώστε να φανεί ότι οι περισσότερες χώρες δωρητές ε, είναι, δεσμεύονται δεσμεύονται και ακόμα πιο σημαντικό είναι η ε, δέσμευση για να βρούμε μια διακυβέρνηση πέρα δηλαδή από το γεγονός ότι ε, θα συμπεριλαμβάνονται όλοι, αλλά θα υπάρχει μια διακυβέρνηση ε, λαφριά σε επίπεδο κάθε ε, χώρας δικαιούχου. Και αυτό ήταν ο ρόλος του UNDP. Για την ώρα θα πρέπει να σας πω ότι διαπιστώνουμε αδυναμίες στην εφαρμογή τοπικό επίπεδο. Υπάρχουν ιδέες για βελτίωση της διακυβέρνησης αυτής. Μία από αυτές τις ιδέες είναι η καλύτερη ενσωμάτωση της εργασίας ε, ε, όσον αφορά το building blocks που εργάστηκαν πριν από τον Μπουσέντρα, πολύ θετική η εξέλιξη και έγιναν και εργασίες παρακολούθησης, ε, πράγμα που δεν είχε γίνει μέχρι στιγμής. Υπάρχουν ιδέες επίσης για να δοθεί πιο σημαντικός ρόλος στις ε, τοπικές ε, αρχές, ώστε να στηριχθεί η Επιτροπή παρακολούθηση, αλλά να υπάρξει και παρακολούθηση όσον αφορά την εφαρμογή σε κάθε χώρα. Υπάρχουν λοιπόν ιδέε για βελτίωση τη διακυβέρνηση, αλλά διαπιστώθηκε ότι για την ώρα υπάρχουν σημαντικέ αδυναμίε και σε αυτό οφείλεται το γεγονός ότι η έκθεση που θα συζητηθεί στο Μεξικό για την παρακολούθηση όλων των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν στο Μπουσάν δεν είναι ακόμα έτοιμη. Και θα είναι έτοιμη μόνο την επόμενη εβδομάδα, πράγμα το οποίο με εμποδίζει να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες. Νομίζω λοιπόν πως στο Μεξικό θα μπορέσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξουμε και κάνουμε μια έκθεση αυτή τη στιγμή με τα κράτη-μέλη μας για τα όσα κάναμε για να θέσουμε σε εφαρμογή τις δεσμεύσεις του Μπουσάν και όχι μόνο του Μπουσάν αλλά και των άλλων ε, προηγούμενων δεσμεύσεων. Ε, την πρόοδο που έχουμε σημα... Ε, επιτύχει όσον αφορά το συντονισμό των στόχων μας ε, για, εδώ και τρία χρόνια για τον κοινό προγραμματισμό με τα κράτη-μέλη μας. Ένα δεύτερο ισχυρό μας σημείο για την Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή και αυτό θα το παρουσιάσουμε στο Μεξικό επίσης είναι η πρόοδος όσον αφορά τη διαφάνεια. Και θα υπάρχουν και άλλες πτυχές που αναφέρονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, αλλά πιστεύω ότι η διαφάνεια και ο κοινό προγραμματισμός, ο συντονισμό είναι τα δυνατά σημεία της Ένωση. όπου έχουμε κάνει δηλαδή τη μεγαλύτερη πρόοδο από το Μπουσάν. Τελευταία παρατήρηση είναι ότι βεβαίω αυτή η διάσκεψη είναι σημαντική, το έλεγα στην αρχή, για την αξιοπιστία της ε, σύμπραξη. Δεν είναι μια διάσκεψη όπου θα εξαγγείλουμε νέε υποσχέσει, αλλά όπου πρέπει να αποδείξουμε ότι έχουμε επιτύχει πρόοδους από τον Μπουσάν και αυτό είναι επίσης σημαντικό διότι προβλέπονται συζητήσεις στον ΟΗΕ για τους μελλοντικούς στόχους που θα αντικαταστήσουν μετά από το 2015 τους στόχους της χιλιετίας. Δεδομένου ότι βλέπουμε την σύμπραξη του Μποσάν ως μια πλατφόρμα που στόχο έχει να σταθεί ενώπιον της διεθνούς κοινότητας ως ε, μια πλατφόρμα εφαρμογής των στόχων που θα αποφασιστούν το Σεπτέμβριο του 2015. Για να μπορέσει λοιπόν το Μπουσάν να παίξει αυτό το ρόλο του πώς θα εφαρμοστούν οι στόχοι μετά το 2015, πρέπει καταρχήν να μπορέσουμε να δείξουμε πως είναι μια σύμπραξη που λειτουργεί, και όπου η δέσμευση όλων των παραγόντων αρκεί ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τις υποσχέσεις μας. Σας ευχαριστώ και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και δίνω το λόγο στην κυρία Σοφία Μπορνόλη από την Business Europe για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολύ χαιρόμαστε που βρισκόμαστε εδώ από την Business Europe για να μοιραστούμε μαζί σας τις απόψεις μας για το πώς ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να βοηθήσει. Τι θέλει, τι θέλει, μπορεί. Για εμάς ε, βεβαίως το... το βασικότερο εδώ πέρα είναι το ότι μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο ο ιδιωτικό τομέα με την ατζέντα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί πράγματι θεωρούν πω πρέπει να υπάρξει περισσότερο χώρο για τον ιδιωτικό τομέα στην ε, διαδικασία διαμόρφωσης ε, της πολιτικής, ειδικά όσον αφορά την καλύτερη μόχλευση των πόρων του ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη. Και βεβαίως έτσι θα μπορούσε να δημιουργηθούν καταστάσεις ε, αμοιβαία επωφελής και για τις αναψώμενε χώρες που χρειάζονται αυτή την στήριξη και για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των ευρωπαϊκών και των τοπικών επιχειρήσεων και αυτό μπορεί να γίνει παραδείγματος χάρη μέσω των ΣΔΙΤ με την συμμετοχή διαφόρων ενδιαφερομένων. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιωτικού τομέα, ειδικά μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και δημοσίων φορέων και μικείο. έτσι ο ιδιωτικός τομέας αφενός ξεκινάει με κάποιες ε, αναπτυξιακές ε, πρωτοβουλίες οι οποίες από την άλλη υποστηρίζονται σε τοπικό επίπεδο μέσω των αναγκαίων εγγύσεων. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες ε, μπορούν να μοιραστούν τις πολύτιμες εμπειρίες τους στις εμπειρίες αυτές. Ε, το έχουν κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια με πολύ σημαντικές πολιτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι πως όταν μια ευρωπαϊκή εταιρεία αποφασίζει να επενδύσει σε μια αναψώμενη χώρα, ένα δίκτυο τοπικών ε, παρόχων, ειδικά μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ε, δημιουργείται και αυτό βέβαια έχει θετικές εξωτερικές επιπτώσεις για τις τοπικές κοινότητες. Για να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Μια εταιρεία ε, ευρωπαϊκή έχει δημιουργήσει ε, μια εταιρεία για την ε, παροχή των βασικών δημητριακών στην Τανζανία. Βοηθάνε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχουν κάποια εργαστήρια εκπαιδευτικά και ο στόχος του έργου είναι να βοηθήσουν τις τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να επεκτείνουν τα προϊόντα τους, να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά και το, μια άλλη ευρωπαϊκή εταιρεία επίσης έχει ξεκινήσει ένα πιλωτικό πρόγραμμα για την βιώσιμη παραγωγή τσαγιού στην Κένια με στόχο τη βελτίωση της ε, παραγωγικότητας, ε, την καλή διαχείριση της ενέργειας, την ε, διαφύλαξη της των τοπικών βιοτόπων. Ήδη έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα, έχει βοηθήσει να αυξηθεί το εισόδημα των αγροτών και βέβαια έχει αυξήσει την τοπική απασχόληση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πρώτα απ' όλα οι ευρωπαϊκοί, ε, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να μπορούν να συνεργάζονται καλύτερα, όπως επίσης βεβαίως και να υπάρξει καλύτερη διοργανική συνεργασία μεταξύ Κομισιών, Ευρωπαϊκής ε, Τράπεζας Επενδύσεων και των διαφόρων κλάδων. Για να δώσω ένα πιο συγκεκριμένο παράδειγμα, εμείς θεωρούμε στην Business Europe πως η πολιτική εμπορίου και ανάπτυξης σχετίζονται και αν σχεδιαστούν σωστά είναι συμπληρωματικές. Οπότε το εμπόριο και οι επενδύσεις ως ένα μέρος ισορροπημένης ε, πολιτικής ε, ανάπτυξης νομίζω μπορεί να βελτιώσουν και την διαχείριση στις ε, χώρες οι οποίες έχουν χαμηλούς πόρους, λίγους πόρους και να βοηθήσουν στη μείωση της στόχης. Κατόπιν, οι διπλωματικές προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο ΟΗΕ και ΟΣΑ. Ε, επίσης και το υψηλό το υψηλού επίπεδου φόρουμ στο Μεξικό είναι μια ιδανική ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να στείλει το μήνυμα στους εταίρους μας, σαν ψώμενες χώρες, πως η αποτελεσματική διακυβέρνηση και το σαφές επιχειρηματικό πλαίσιο έχει μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη και επίσης θα βοηθήσουν στην προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων. Αυτό είναι ο ρόλος μας ως ε, εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα. Θα είμαι σύντομη. Ναι. Θα ήθελα να καταλήξω με το εξή για εμά είναι σαφές πως ο ιδιωτικός τομέας έχει να παίξει ένα ρόλο στην ανάπτυξη. Είναι επίσης σαφές πως ε, η προσέγγιση αυτή μοιάζει να είναι πιο αποτελεσματική στον ε, τομέα αυτόν καθώς ε, εδώ πέρα έχουμε καλύτερη μόχλευση των πόρων, των χρημάτων δηλαδή στην ανάπτυξη και ταυτόχρονα διασφαλίζεται πως το όφελος μένει στην τοπική κοινωνία. Σας ευχαριστώ και αναμένω τις ε, τυχόν ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole. Ευχαριστούμε. Τώρα, το λόγο έχει η κυρία Σουζάννα Σκάντοβα, που είναι από το Κονκόρτ. Τέσσερα λεπτά κι εσείς, επειδή έχουμε καθυστερήσει πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε και εμείς που μας καλέσατε στη συζήτηση αυτή που αποτελεί στοιχείο κλειδί για το μέλλον θα σας παρουσιάσουμε τις ε, απόψεις μας για την διαδικασία αυτή. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό για τις ε, οικονομικές εξελίξεις και για το πλαίσιο μετά το 2015. Η αποτελεσματικότητα της ενίσχυσης έχει ξεκινήσει από το 2002 που αναγνωρίσαμε όχι μόνο ποσοτικά μέτρα αλλά και ποιοτική βοήθεια. Από τότε έχουν λάβει χώρα διάφορα φόρα στη Ρώμη, το Παρίσι, Μπουσάν κλπ. Και στο Μπουσάν, για παράδειγμα, το 2011 το θέμα της αποτελεσματικότητας της ενίσχυσης οδήγησε σε μια νέα εταιρική σχέση με τη φιλοδοξία να ακούγονται οι φωνές όλων των ε, εμπλεκομένων. Η συνεργασία λοιπόν άλλαξε και περάσαμε από την ενίσχυση στην αποτελεσματικότητα. Κάτι με το οποίο είχαν συμφωνήσει οι εταίροι και στο Παρίσι και στην Άκρα. Σε δύο χρόνια λοιπόν μετά το Μπουζάν η αποτελεσματικότητα της ενίσχυσης αποτελεί πολύ σημαντικό μέρος της ατζέντα και όντως πρέπει να ενισχυθεί ακόμα η αρχή αυτή. Η πρώτη συνάντηση των εταίρων στο Μεξικό θα καθορίσει το μέλλον τη ατζέντα για την αποτελεσματικότητα της ενίσχυσης. Η συνάντηση αυτή πρέπει να αντικατοπτρίζει και την πρόοδο που επιτυχάνεται μετά το Μπουσάν που έγινε πριν από δύο χρόνια, αλλά και να εντοπίσει μέτρα ώστε να πάψουν να υπάρχουν τα εμπόδια που υπάρχουν σήμερα. Το Μεξικό λοιπόν θα είναι μια ευκαιρία για να αξιολογήσουμε την συμμετοχή, τα αποτελέσματα του Μπουσάν, ε, αξιολόγηση της εντολής και γενικότερα τις εταιρικές σχέσεις. Στα πλαίσια άλλων ε, σημαντικών ε, στοιχείων και εν ώψη του 2015 που είναι ο στόχος μας, το Μεξικό αποτελεί μια ευκαιρία για να αλλάξει τάση και η αποτελεσματικότητα της ενίσχυσης να πετύχει. Κυρίως μετά τις εξελίξεις μετά το 2015 η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι από τους μεγαλύτερους δωρητές, πρέπει να παίξει ρόλο κλειδί και να αποτελέσει το παράδειγμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες μέλη πρέπει να αποφασίσουν για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα μετά το Μεξικό και να διασφαλίσουν ότι το Μεξικό θα φέρει αποτελέσματα για περισσότερη συμμετοχή στην ανάπτυξη. Βέβαια πρέπει να προβληματιστούμε στα πλαίσια του διετούς προγράμματος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Επιτροπή κάνει μια μελέτη για την πρόοδο όσον αφορά τις υποχρεώσεις που αναλάβαμε στο Μπουζάν, αλλά πιστεύουμε ότι χρειάζεται συνεχής εποπτεία μέσω της έκθεσης λογοδοσίας, για παράδειγμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προχωρήσει περισσότερο και στην πολιτική της για να βρεθεί πιο κοντά σε αυτούς που έχουν ανάγκη για να αντιμετωπίσει τις ανισότητες, να βοηθήσει τους πιο ευάλωτους μέσω συνεργασίας και πολιτικού διαλόγου με όλες τις χώρες. Και για να είναι αποτελεσματική πρέπει να λάβει υπόψη της την απάλληψη της ένδυας, να ενισχύσει τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι νέοι δωρητέ αποκτούν όλο και μεγαλύτερη αξία, όπως και η περιφερειακή συνεργασία, και αυτό και ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει ρόλο διευκόλυνσης, καταλητικό και να ενισχύσει την τριμερή συνεργασία στις διαφορε περιφέρειες. Πιστεύουμε ότι ο ιδιωτικό τομέα έχει να παίξει πολύ θετικό ρόλο, αλλά και αρνητικό μερικές φορές. Γι' αυτό και χρειάζεται πολύ συγκεκριμένη αξιολόγηση για το τι μπορεί να προσφέρει συμπληρωματικά και για να στηρίξει τους αναπτυξιακούς στόχους. Η αποτελεσματικότητα της ενίσχυσης είναι η απάντηση στην συνεργασία. Μετά το 2015 τι ακριβώς θα σημαίνει αυτό πρέπει να υπάρχουν αποτελέσματα. Γι' αυτό χρειάζεται ένα πλαίσιο για την αναπτυξιακή συνεργασία που να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της εποχής μετά το 2015. Συνεπώς, το αναπτυξιακό πλαίσιο μετά το 2015 πρέπει να προϋποθέτει την δέσμευση, τη διαφάνεια, την λογοδοσία, αποτελέσματα, συμμετοχή όλων και αποτελεσματικότητα της ενίσχυσης στο Μεξικό και μετά το Μεξικό οι συμπρόεδροι, οι υπουργοί, τα μέλη του steering group κλπ. πρέπει να δεσμευτούν στις αρχές αυτές και να συμπεριληφθούν σε ένα πλαίσιο για μετά το 2015 αναγνωρίζοντας τη δουλειά μένει να γίνει ακόμα για να βελτιωθεί η πρακτική μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γκέρενς έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Οι διάφορες διασκέψεις που αναφέρθηκαν στη συζήτηση εδώ, στις παρεμβάσεις που ακούσαμε, μας υπενθυμίζουν Μόντερε, Μπουζάν, Μπαλί, Άκρα. Αυτό επιβεβαιώνει ότι υπάρχει ένα πολυμερές πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνεται η συζήτησή μας. Να το ξέρουμε αυτό, ότι συμμετέχει η διεθνής κοινότητα και πρέπει να παραμείνει αυτό το διεθνέ πλαίσιο. Δεύτερο, τι θετικό μπορούμε να κάνουμε στο Μεξικό και ποιο είναι αυτός που θα κάνει τη διαφορά. Έχοντα ακούσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία πολύ σωστά λέει ότι δεν θέλει να φύγει μάδια τα χέρια, πρέπει να στοιχηματίσουμε ακριβώς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου εκείνη να θέσει νέα ζητήματα με το βάρος που έχει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, δεν ξέρω ποιος τελικά θα εκπροσωπεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα πρέπει να είναι μετριόφρον εκεί. Αντίθετα, έχουμε πραγματονομοσύνη να φέρουμε. Και είναι και ένα μάθημα που έχω πάρει από δύο συναντήσεις στα πλαίσια του διαρθρωμένου διαλόγου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποιος έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη. Εγώ επέμεινα στη διάσκεψη του Μοντερή, ήταν ακόμα η διεθνής κοινότητα που δεν έκανε αρκετές προσπάθειες για να χρηματοδοτήσει την αναπτυξιακή προσπάθεια. Και όλοι ορκίστηκαν για το 0,7% παρόλα αυτά δεν το πετυχαίνουμε, ούτε το 0,5% δεν καταφέρνουμε. Συνεπώς, είναι και θέμα διαπαιδαγώγησης. Αν υπενθυμίζουμε τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει, ίσως κάποτε τα καταφέρουμε. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύω ότι ακριβώς πρέπει να επιμείνει για την αλλαγή. Αν πραγματικά δεν θέλουμε αρνητικό απολογισμό ξανά. Όσον αφορά την εκπλήρωση των στόχων της χιλιετίας για την ανάπτυξη, πρέπει να επιμείνουμε στην ευθύνη που έχει κάθε χώρα. Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι πραγματικά μια κρίση σε όλες τις χώρες. Στις αναδυόμενες χώρες δεν συζητάνε τίποτα άλλο πέρα από τη μείωση των ανισοτήτων. Και ποιος θέει. μα ίδιες οι χώρες. Όταν παράγουν πλούτο πρέπει να τους το πούμε και πρέπει να επιμείνουμε ακόμα περισσότερο στις χώρες που το χρειάζονται πιο πολύ. Συνεπώς πρέπει να τονίσουμε την διαφοροποίηση αυτή. Η διαφοροποίηση δεν σημαίνει ότι ξεφεύγουμε από τις ευθύνες μας, Απλώς μεταφέρουμε τις ευθύνες μας στους άλλους. Συνεπώς, να φανεί φιλόδοξη στο Μεξικό η Κομισιόν και να βάλει όλους τους υπεύθυνου απέναντι στις ευθύνες τους. Όσοι δεν έχουν ακολουθήσει την Κομισιόν θα πρέπει να στηθούν από την Κομισιόν στον τοίχο. Ευχαριστούμε πολύ, Λή Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συνομιλητές μας για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Ερχόμαστε τώρα στο τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης, τα διάφορα πρώτα απ' όλα. Πήραμε επιβεβαίωση ότι η Καθιάστον, η εκπρόσωπος και την πρόεδρος της Επιτροπής θα υπογράψει στις 3 Απριλίου την ε, Συμφωνία για την Ανάπτυξη. Πολλές φορές της το έχουμε ζητήσει γιατί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης πια παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην αναπτυξιακή πολιτική και συνεπώς αυτή η συμφωνία, αυτό το consensus αποτελεί μια πολύ καλή βάση για την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κάτι που έχουν συντάξει από κοινού η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και έχει συνεπογραφεί από τους τρεις Προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήδη από το 2005. Είναι πολύ καλό νέο λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης μέσω της ΥΠΑ του εκπροσώπου συνυπογράφει επίσης το κείμενο αυτό σε μία εκδήλωση την οποία οργανώνει ο πρόεδρος Σούλτς. Παρακαλώ κύριε Γκέρεντς. Ευχαριστώ πολύ, έτσι πολύ όμορφα θα τελειώσει η θητεία αυτή. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να συμβιβάσουμε τις φιλοδοξίες της Επιτροπής μας. Χαίρομαι πολύ που τελικά δέχτηκε η Λέιντι Άστον την αρχή της υπογραφής αυτής και που τήρησε την υπόσχεσή της. Ήταν ε, υπόσχεση που έδωσε σε μια συνάντηση που είχαμε δώσει αυτή την ίδια την αίθουσα. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή για το Κοινοβούλιο. Δώσαμε αγώνα για να το πετύχουμε. Όλα καλά εφόσον τελειώνουν καλά. Ωραία. Δεν μένει παρά να σας ανακοινώσω την προσεχή μας συνεδρίαση. Στις Βρυξέλλες, την 3η 1η Απριλίου, 9 με 12 και 30, και την Δευτέρα 7 Απριλίου, που θα είναι και η τελευταία συνεδρίασή μας, 3 με 6.30